για να, ένα αίτημα για να γίνει μια μελέτη θελήσαμε να έχουμε μια ε, εποπτεία με γενική εικόνα ε, του κατά πόσο να κράτη-μέλη ε, τηρούν το πρόγραμμα Natura 2000 και να μπορούμε να γνωρίζουμε τι πρέπει να συμπεριληφθεί στο μέλλον στην μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και έχει διανεμηθεί στα μέλη μέχρι τώρα μόνο στα αγγλικά. Ε, όπως είχαμε στήσει, εντοπίζονται τα βασικά θέματα ανάμεσα στην ε, Natura 2000 αλία, περιγράφει την όλη διαδικασία και την ε, εφαρμογή, αλλά όπως και τις διάφορες λύσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τον συντάκτη αυτής της έκθεσης, τον κύριο Χάνε Φοκ από το Αμβούργο, που θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση για τα βασικά πορίσματα της έκθεσής του και κατόπιν μπορούμε βέβαια να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι, κύριε Φοκ. αυτή η οθόνη πάνω από το κεφάλι μου, λέει ο Πρόεδρος, ε, δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο. Γι' αυτό θα πρέπει να στρέψετε το βλέμμα σας ε, στις άλλες δύο ε, οθόνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου προσφέρετε η ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτό το θέμα που είναι το Natura 2000 και η κοινή ελληνική πολιτική. Σήμερα το απόγευμα θα εστιάσω την προσοχή μου σε βασικές ε, ανάγκες ε, που υπάρχουν όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος 2000 ε, και πάντα σε σχέση με την κοινή ελληνική πολιτική. Θα εστιάσω την προσοχή μου σε βασικά θέματα της κοινή ελληνική πολιτικής και της Natura 2000, πώς αυτά τα θέματα σχετίζονται μεταξύ τους. Κατόπιν θα αναφερθώ σε κάποια θέματα πολιτικής που είναι πολύ σημαντικό να γίνουν κατανοητά και μετά θα σας επισημάνω τέσσερα ε, θεμελιώδη θέματα, τα οποία ίσως μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της κοινή ελληνικής πολιτικής του μέλλοντος. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να πούμε για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ε, αυτή είναι μια βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, την πολιτική τη διαχειρίζονται ε, κυρίως η Επιτροπή και τώρα και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι να αναζητήσει τους φυσικούς πόρους με βιωσιμότητα ε, επίσης να εντοπίσει οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Όσον αφορά τους βιότοπους ε, του Natura 2000, έχουμε τον κανονισμό του Συμβουλίου του 92 που περιγράφει το στόχο και ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιοπικιλότητα μέσα από τη διατήρηση των φυσικών βιοτόπων και της άγριας κλωρίδας και πανίδας. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο το πρόγραμμα Natura 2000 είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων, θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και είναι ένα εργαλείο της οδηγίας περιβιοτόπων, ένα εργαλείο για να επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν είναι ε, οι βιότοποι και τα είδη που αναφέρονται σε διάφορα παραρτήματα της σχετικής οδηγίας να διαφυλαχθούν και επ' αυτού θα επανέλθω αργότερα. μετά τη μεταρρύθμιση του 2003 της κοινή ελεκτικής πολιτικής ε, έλαβε χώρα, ξεκίνησε μάλλον, μια δεύτερη μεταρρύθμιση πρόσφατα και η συζήτηση ξεκίνησε το 2009 σχετικά με τη μεταρρύθμιση. Στόχοι αυτής της ε, μεταρρύθμισης της κοινή ελεκτικής πολιτικής στο μέλλον, οι στόχοι διαχωρίζονται σε δέκα διαφορετικά θέματα και ένα εξ αυτών είναι το ε, διαφοροποιημένο καθεστώς διαχείρισης που σημαίνει ότι έχει ως ε, στόχο διαφοροποιημένη διαχείριση, εντοπισμό της παράκτιας αλίας, ε, εντοπισμός της αλίας ανοιχτού πελάγους και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε την περιφερειοποιημένη διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο θέμα της μελλοντικής πολιτικής, της αλληλευτικής, ε, είναι να υπάρχει η περίφημη έννοια του MSI, Maximum Sustainable Yield. Δηλαδή, να υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα από την αλία και αυτό να οδηγήσει στη μείωση των προσπαθειών αλίας. Ένα άλλο θέμα είναι να ενισχυθεί η παράκτια αλία, να ε, ενισχυθεί, να υποστηριχθεί η αλία των απλών ψαράδων και επίσης και να ε, ενισχυθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Τέλος, θα ήθελα να εξετάσω και το μέλλον της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ότι αυτή πρέπει να είναι τμήμα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε το πώς η κοινή αυτή πολιτική μπορεί να προσφέρει τα σωστά εργαλεία για να στηρίξουμε το οικοσύστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που η κοινή αλληλευτική ε, πολιτική ε, θα προσπαθήσει να ε, αντιμετωπίσει και να συστήσει μέσω αυτών το οικοσύστημα. Η οδηγία περί βιοτόπων, όπως σας ανέφερα, δημοσιεύθηκε το 1992 και έκτοτε έχουν λάβει χώρα πολλές εξελίξεις. Η κοινή αλληλευτική πολιτική ξεκίνησε το 1984, έχει λοιπόν να επιδείξει μια μακρά αλλαγή, μακρά ιστορία αλλαγών και προσαρμογών. Ε, το 1992 είχαμε για πρώτη φορά την έννοια της, ε, του οικοσυστήματος και την έννοια της ε, βιώσιμης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Το 1992 δημοσιεύτηκε η οδηγία περί βιοτόπων και τα πρώτα χρόνια η οδηγία αυτή είχε ε, σχέση με τα θαλάσσια οικοσυστήματα της ανοιχτής ε, θάλασσας. Δεν έγιναν και πολλά πράγματα έκτοτε. Ε, το 2005 αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη πέρα από τα 12 μίλια. Στον τομέα αυτό ε, πράγματι υπήρξε κάποια πρόοδος. Κατόπιν το 2007 η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δημοσιεύθηκε με στόχο να συμπεριλάβει όλες ε, τις ε, θαλάσσιες πολιτικές κάτω από μια ομπρέλα με ευρύτερο απότερο στόχο στον τομέα αυτό να συντονιστούν όλες οι πολιτικές για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον και εν ευθέτω χρόνο να υπάρξει συντονισμός και με το ε, πλαίσιο το οποίο καθορίζει η οδηγία και το οποίο δημοσιεύθηκε με περισσότερο οικολογική απόχρωση έχοντας ως στόχο να επιτευχθεί προστασία του περιβάλλοντος, ε, κυρίως όσον αφορά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα υδρόβια οικοσυστήματα. Πέρα από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε και περιφερειακά πλαίσια που καταρτίστηκαν και αυτά, όπως παραδείγματος στην Επιτροπή ΟΣΠΑΡ στο Παρίσι το 2003. Ε, μία έννοια ενός ε, της προστατευόμενης ε, θαλάσσιας πολιτικής, αυτή συμβάδισε ε, με την οδηγία περί τόπων. Και το 2010, στην εφετινή συνάντηση των Υπουργών, η ΟΣΠΑΡ άρχισε να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για να συμπεριλάβει όλες τις ε, θαλάσσιες πολιτικές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από μια ευρύτερη ομπρέλα και με τον τρόπο αυτό να ενσωματωθούν η θαλάσσια στρατηγική, η Natura 2000 και θέματα λίας. Όλα αυτά να ενταχθούν σε μία και μόνο πολιτική. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και η εξέλιξη των διαφόρων πολιτικών τα στοιχεία είναι αρκετά περίπλοκα. Αριστερά βλέπουμε ότι η κοινή ελευτική πολιτική είναι θεμελιώδης αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή εξετάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αλία πέρα από τα 12 ναυτικά μίλια και επίσης και στα παράκτια ύδατα στο βαθμό που βέβαια τα κράτη-μέλη ε, έχουν παραχωρήσει την πρόσβαση σε αυτά τα ύδατα μέσα από διεθνείς ε, συμφωνίες που ενδεχομένως έχουν ε, συναυθεί. Κατά τα άλλα, βλέπετε αυτό που είναι η EZ, αυτή είναι η πλήρης αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν οτιδήποτε έχει σχέση με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων όπως είναι το πετρέλαιο, το αέριο, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, εδώ παίζουν ρόλο και τα θέματα της προστασίας της φύσης. Όσον αφορά τώρα στην οδηγία για το θαλάσσιο πλαίσιο και την Natura 2000, τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα αλλά και την αρμοδιότητα να καταρτήσουν προγράμματα διαχείρισης. Από τη στιγμή βέβαια που επηρεάζεται η αλία, αυτά τα προγράμματα διαχείρισης πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αποτελούν τμήμα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ενώ προγράμματα διαχείρισης που έχουν σχέση με άλλους χρήστες, αυτά μπορούν να εκπονούνται και να δημοσιεύονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τώρα το ολοκληρωμένο θαλάσσιο πλαίσιο. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που σας ανέφερα προηγουμένως και πέρα από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τις ε, θαλάσσιες συμφωνίες όπως είναι η ΟΣΠΑΡ, την ΧΕΛΠΑ για την Βαλτική και ε, τα κράτη-μέλη ορισμένες από τις αρμοδιότητές τους τις μεταφέρουν στην ΟΣΠΑΡ, όπως παραδείγματο χάρη τον ορισμό των περιβαλλοντικών στόχων. ΟΣΠΑΡ, όπως σας είπα προηγουμένως, προσπαθεί να συμπεριλάβει την ε, θαλάσσια πολιτική και τα θέματα της Natura 2000 κάτω από μία και μόνο ομπρέλα. Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε νέα καταληκτική ημερομηνία για τα κράτη-μέλη για να καταρτήσουν τους ε, καταλόγους ε, των ε, χώρων της θαλάσσιας της Natura 2000, θαλάσσιους χώρους της Natura, του Natura 2000 αυτού του προγράμματος. Και αυτά έπρεπε να γίνουν στο χρονικό πλαίσιο των τριών χώρων. Από τη στιγμή που θα έχουν υποβληθεί αυτοί οι θαλάσσιοι χώροι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τις προτάσεις και μετά από την έγκριση αυτών των χώρων ε, θα περάσουν άλλα εξι χρόνια η οποία ως περίοδος προσφέρεται για τα κρατημέλη για να αρχίσουν να προετοιμάζουν ε, μέτρα διαχείρισης αυτών των χώρων, να προετοιμάσουν τα προγράμματά τους ε, όσον αφορά στην αλία. Και αυτά τα προγράμματα να υποβληθούν και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές για το 2007 για να υπάρχουν προστατευόμενοι θαλάσσιοι χώροι. Σχεδιάστηκαν και ορίστηκαν οι χώροι αυτοί. Και το 2008 δημοσιεύθηκε το έγγραφο αυτό το οποίο περιλάμβανε για τα κράτη-μέλη έναν κατάλογο ε, έτσι ώστε να προετοιμάσουν ε, προγράμματα διαχείρισης. Ε, κατ' ουσίαν κανένα κράτος μέλος δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και υπάρχουν κάποια προγράμματα άλλα διαχείριση, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της εξέλιξης. Όσον αφορά σε αυτόν τον κατάλογο θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν πριν υποβληθούν τα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν τέσσερα θέματα τα οποία δεν είναι ακόμα όριμα από πλευράς ε, μεθοδολογίας. Δηλαδή, πρώτον, πώς να εντοπίζονται οι απειλές στους βιότοπους, ε, πώς να γίνεται κατά δεύτερον η διαφοροποίηση των διαφόρων αλληλευτικών πολιτικών, ε, πώς να συμπεριλαμβάνονται οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή τη διαδικασία της κατάρτισης προγραμμάτων διαχείρισης, πώς να συντονίζονται τα πράγματα που αφορούν στην προστασία της φύσης ε, με ε, διασυνοριακά, διασυνοριακούς βιότοπους. Πώς να αντιμετωπιστούν θέματα μετατόπισης. Δηλαδή όταν η αλία αποκλείεται από ένα συγκεκριμένο χώρο, τότε πρέπει να μεταφερθεί σε έναν άλλο χώρο που να είναι απόλυτα προσπελάσιμος. Και αυτό βέβαια προκαλεί κάποιες επιπτώσεις, τις επιπτώσεις ε, μετατόπισης όπως αποκαλούνται. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αυτά τα τέσσερα θέματα, αν τα δει κανείς κάπως γενικότερα, καταλήγει, ε, εγώ τουλάχιστον κατέληξα, σε τέσσερα θέματα κλειδί που έχουν σχέση με την κοινή πολιτική και το πρόγραμμα Natura 2000. Το πρώτο θέμα είναι ε, μία στάνταρτ περιγραφή των επιπτώσεων, έτσι ώστε ε, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα. Το δεύτερο είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα κυριότητας. Αυτό έχει σχέση με την μετατόπιση. Ε, πώς μπορούμε να ορίσουμε τα, τις στάνταρτ διαδικασίες για να συμπεριλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι καθότι κάθε έξι χρόνια η διαχείριση πρέπει να αναθεωρείται αφού βεβαίως ε, λαμβάνει χώρα. Και τέλος, πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα δύο συναριακά θέματα. Επ' αυτού θα σας παρουσιάσω κάποια παραδείγματα στο βαθμό που υπάρχουν. Όπως ε, σας είπα, εδώ έχουμε να κάνουμε με πρόοδο. Ε, βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα τα τελικά προγράμματα προς ανάλυση. Όσον αφορά την στάνταρτ ποσοτική περιγραφή των επιπτώσεων. Εδώ χρειαζόμαστε μια εξειδικευμένη ανάλυση έτσι ώστε αυτή να συνδυαστεί με τις προσπάθειες που καταβάλλονται και αυτό εντάσσεται ε, στο πρόγραμμα ελέγχου ε, της αλίας. Αυτό το πρόγραμμα δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη μας τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, την ε, προχωρημένη τεχνολογία και να μπορούμε και να αναλύουμε ε, αντισταθμίσεις. Δηλαδή, όταν περιορίζουμε τις επιπτώσεις ε, μιας συγκεκριμένη εξέλιξης, είναι πολύ πιθανόν ότι οι αλληλείς θα μεταφερθούν σε έναν άλλο τομέα, όπου εκεί βέβαια θα υπάρχουν άλλες ειδικέ επιπτώσεις Ίσως ε, μπορεί κανείς να σκεφτεί ε, το να αντικαταστήσει το bottom gear με το specific gear. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση θα πρέπει να είναι δυνατόν να αναλυθεί. Μία λύση είναι και αυτή εφαρμόζεται πειραματικά στη Γερμανία η εφαρμογή ενός ε, μοντέλου ανάλυσης κινδύνων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια αποτίμηση των κινδύνων και αποκτούμε μια ποσοτική εικόνα του τι ακριβώς ε, λαμβάνει η χώρα. Λυπάμαι που δεν μπορείτε να διαβάσετε καλά αυτό το γράφημα, αλλά έχουμε τέσσερα Έχουμε στις στήλες, ε, τις διάφορες κοινότητες, που περιλαμβάνουν ε, στοιχεία οικοσύστημάτων και έτσι μπορούμε να δούμε ε, ποιο οικοσύστημα τα πηγαίνει καλά, έχει καλή απόδοση. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να έχουμε περιορισμένη αναφορά. Αυτό το βλέπετε με τις τελίτσες που υπάρχουν στο γράφημα. Ε, και κατόπιν μπορούμε να αρχίσουμε να ορίζουμε στόχους για τις ε, διάφορες πολιτικές. Αυτό είναι τμήμα της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσιας ε, προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να εξετάσουμε ειδικέ ρήτρε που αφορούν στην θαλάσσια πολιτική. Μπορούμε να δούμε την έννοια της μέγιστης απόδοσης. Υπάρχουν διάφορα σενάρια και αυτά όλα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Γιατί σε πάρα πολλούς δείκτες ε, βλέπουμε ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Εξάλλου μπορούμε να εξετάσουμε και τις ανάγκες της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Μπορούμε να δούμε το θέμα της ε, περιφερειοποίησης ε, που και αυτό εντάσσεται στην μελλοντική έννοια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Βλέπουμε ότι όλα αυτά τα θέματα ορίζονται και με βιογραφικές μονάδες. Έχουμε δηλαδή το θέμα της περιφέρειας, της, ε, του πληθυσμού, το δημογραφικό. Γνωρίζουμε το κομμάτι του πληθυσμού που επηρεάζεται. Επίσης ε, έχουμε ειδικέ ε, απαντήσεις ε, για το πρόγραμμα Natura 2000. Μπορούμε να δούμε αυτά που αναφέρονται εδώ με πράσινο βελάκι. Μπορούμε να δούμε και τα οικοσυστήματα που αποτελούν τμήμα των ε, υδροβιότοπων που πρέπει να προστατευθούν. Επίσης, μπορούμε να δούμε ε, κατά να έχει επιτευχθεί το ευκταίο επίπεδο προστασίας. Μπορούμε να αναλύσουμε τους, ε, τις ε, απειλές και με τον τρόπο αυτό μπορούμε τελικά να δούμε ε, πώς τα οικοσυστήματα με πιο διαφορετικούς τρόπους. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να εντάξουμε στην ε, κοινή ελευτική πολιτική, στις ε, θαλάσσιες πολιτικές, γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν στην κοινή ελευτική πολιτική όχι μόνο οι προτάσεις του προγράμματος Natura 2000, αλλά να δούμε και πώς η κοινή ελευτική πολιτική μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβάνουν διαφορετικούς στόχους. Το δεύτερο βασικό ζήτημα το οποίο ανέφερα ήταν ε, οι χωροταξικές ιδιότητες των ψαριών. Ξέρουμε την κατανομή ε, των ε, ψαριών και εδώ αυτή είναι μια κοινή ε, πολιτική για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι τάσεις και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί η βιώσιμη ελεία. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τα, τα ψάρια σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πλέον δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Η λίστα μπορούσε να είναι να ορίσουμε τις βασικές ε, ζώνες για την αλία και να τα συμπεριλάβουμε στον χωροταξικό σχεδιασμό ε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι τρόπο ε, να έχουμε ολοκληρωμένε θαλάσσιε πολιτικέ. Στόχο είναι. Στόχος είναι η ίδια η στόχη τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερική πολιτική του 2010. Ε, η πρόσβαση στην παράκτη αλία, η περιφερειοποίηση. Υπάρχει περιφερειοποιημένη αλία. Για παράδειγμα, σας αναφέρω την Ολλανδία, Δανία και τη Γερμανία, ε, τα τμήματα αυτών των χωρών στην Ανατολική Βόρεια Θάλασσα για τα μικρά πελαγικά είδη και κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύουμε τις απειλές ε, μέσα στο χώρο και να βλέπουμε την επίπτωση της μετακίνησης, άπως και καταλάβουμε την συμπεριφορά των ψαριών στο χώρο. Όσον αφορά την παράκτη αλία, να ε, επιστήσω την προσοχή σας στο, ε, στο σχήμα στα δεξιά. Εδώ βλέπουμε αυτές τις προβλεπόμενες, ε, τις προβλεπόμενες ζώνες ε, όπου υπάρχουν νεολικά πάρκα και όπου δεν θα επιτρέπεται η ε, ελίες στις περιοχές αυτές. Μετά με το πράσινο έχουμε το Natura 2000, τους, όπως ακριβώς έχουν οριστεί τις ζώνες Natura 2000, όπως έχουν οριστεί με βάση από την Επιτροπή. Και αν δούμε αυτό το σενάριο, θα δούμε ότι έχουμε απώλεια 50% ε, ε, ευκαιριών αλίας, κυρίως ε, για τη γλώσσα και τους πλάτακες, για τα επίπεδα ψάρια δηλαδή. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ε, πώς μπορούμε να έχουμε τυποποιημένες διαδικασίες ε, ε, λήψης απόφασης, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις γνώσεις όλων των εμπλεκομένων και θα πρέπει να δούμε τις διαδικασίες και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα δεν είναι σαφές το πώς μπορεί να επιτευχθεί είτε στα πλαίσια του ΆΕΣΑΣ, ε, του Διεθνούς δηλαδή Συμβουλίου για την ε, εξερεύνηση των ε, θαλασσών, τα περιφερειακά ράξ, τα συμβούλια και η Ευρωπαϊκή SCCF. Αυτό είναι ουσιαστικό για να καλύψουμε και τους στόχους με βάση τα οικοσυστήματα που είναι η διατήρηση των ειδών, η περιβαλλοντική στόχη, ουσιαστικό επίσης την περιφερειακή προσέγγιση τη μεταρρύθμιση τη ε, κοινή ελευτική πολιτική και ουσιαστικό για τι κατευθύνσει γραμμέ για να αναπτύξουμε προτάσει για μέτρα και να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Διάφορα σχέδια έχουν αληφθεί μέχρι στιγμή. Το πιο πρόσφατο σχέδιο υλοποιήθηκε από, τις, ε, από την Ολλανδία, ΦΥΜΠΑΣ, fishery management in marine protected areas, ε, διαχείριση αλίας σε θαλάσσια προστατευόμενε ζώνες. Αυτό το φύμπας χαρακτηρίζεται από ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι ο συντονισμός γίνεται από το Εθνικό Υπουργείο πριν ξεκινήσει το σχέδιο, οι εμπλεκόμενοι που είναι οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικέ οργανώσει και οργανώσει αλλιέων συμπεριλήφθηκαν στη διαδικα... συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού. Υπάρχει επίση ε, ε, ε, συμβολή επιστημονική εκ μέρου του ISIS και σε, ακόμα και σε αυτό το τόσο ε, πρώιμο επίπεδο συμπεριλήφθηκε η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Το ΦΥΜΠΑΣ βεβαίω ωφελήθηκε από την εμπειρία άλλων προηγούμενων σχεδίων όπως για παράδειγμα το H.E. Winds, ε, που είχε να κάνει με τις Ιρλανδικές προστατευόμενες ζώνες. Τέλος, εξετάζοντας ε, συνοριακά ζητήματα, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολύ διαφορετικές ε, προσεγγίσεις όσον αφορά τον ορισμό των στόχων διατήρησης. Βλέπουμε την Dogger Bank που είναι στην κεντρική βόρεια θάλασσα, και τις γειτονικές περιοχές. Εδώ ε, τρία διαφορετικά κράτη-μέλη όρισαν ε, πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, ε, πολύ διαφορετικό αριθμό στόχων. Το ζήτημα είναι τώρα το πώς μπορούν όλα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού και ποιο θα αναλάβει το συντονισμό. Άρα, μια λίστα μπορούσε να είναι ένα μέσο ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής ή η μεταφορά του ζητήματος αυτού σε υψηλότερο επίπεδο, όπως και στην περίπτωση του ΟΣΠΑΡ. Αλλά βεβαίως το ΟΣΠΑΡ ε, είναι ανεξάρτητο από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εν είδη συμπεράσματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι Τώρα η Ευρωπαϊκή Ελία αντιμετωπίζει ένα, ένα μεγάλο έυρος νέων περιβαλλοντικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τι διάφορε ε, ευρωπαϊκέ θαλάσσιε πολιτικέ. Είναι οι, οι κότοποι, τα οικοσυστήματα, οι περιβαλλοντικέ πτυχέ τη κοινή ελευθερική πολιτική και επίσης ε, οι συμβάσεις, οι διεθνείς θαλάσσιες συμβάσεις, π.χ. Όσπορ και Έλκομ. Από τότε που ε, η ελληνική πολιτική είναι βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και, ε, και υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία για μια προσέγγιση εκ μέρους των οικοσυστημάτων, η κοινή ελευτική πολιτική θα μπορούσε να παίξει σημαντικό και κεντρικό ρόλο αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε να, ε, να, να διαθέτει τυποποιημένα πρωτόκολλα για την ε, ε, εφαρμογή όλων αυτών των περιβαλλοντικών διαδικασιών και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλο πολιτικό μέσο το οποίο να έχει αυτή την κεντρική ε, αρμοδιότητα παρά μόνο την κοινή ελευτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την τόσο ενδιαφέρουσα σα παρουσίαση. Πρέπει να σα πω, με εξέπληξε όταν άκουσα να λέτε ότι κανένα από τα 27 κράτη-μέλη δεν έχει ολοκληρώσει τα σχέδια διαχείρισης. Δεν θέλω να πω, ε, γιατί έχετε καμιά ιδέα γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτό. Ναι, ε, να σα πω το εξή. Ε, τελείωσαν οι διορισμοί μέχρι το 2008 ή εξακολουθούν ακόμα να βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 2008 στην 6 χρόνια φτάνουμε στο 2014. Απλή υπολογισμοι υπολογισμοί. Ορισμένα κράτη-μέλη Ε, έκαναν τους ορισμούς πολύ νωρίτερα και αυτά τα κρατή όπως η Γερμανία θα πρέπει να έχουν τα σχέδια διαχείρισης μέσα το 2012. Ωραία, μάλιστα. Κύριε Σλόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ήταν πολύ διαφωτιστική η παρουσίαση και μου άρεσε πολύ η εικόνα με όλα αυτά τα πλαίσια της νομοθεσίας και καθώς και τις συμβάσεις πραγματικά είναι πολύπλοκη αυτή η εικόνα και είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε τους ε, στόχους της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων πόρων, εξασφαλίζοντας και τη βιοπικιλότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον ταυτόχρονα. Βράτω με τις ευκαιρίες για να σας δώσω ένα ειδικό παράδειγμα. Δεν υπάρχουν και τόσοι βουλευτές, οπότε μπορώ ίσως να χρησιμοποιήσω λίγα περισσότερα λεπτά. Οι εθνικές αρχές έκαναν το σχεδιασμό όπως έπρεπε σε σχέση με τις θαλάσσιες περιοχές που θα έπρεπε να ενταχθούν στο Natura 2000 στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και τοπίσαν, όπως θα έπρεπε, βέβαια, και τις ε, βασικές απειλές που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον. Η κατάληξη ήταν ότι η μεγαλύτερη απειλή που κατά των προστατευόμενων αυτό, μάλλον των περιοχών που θέλουν να προστατεύσουν, ε, είναι η αλία βυθού με αλληλευτικά εργαλεία σειρώμενα στο βυθό. Πώς μπορούμε, είπαν λοιπόν οι σχετικές αρχές, να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Πρέπει ε, το bottom trolling, αυτό το είδος αλίας, να σπάψει να χρησιμοποιείται και απευθύνθηκαν στο Σουηδικό Συμβούλιο Αλία που είπαν ότι όχι, δεν μπορούμε να σα πούμε τίποτα γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα τη κοινή αλευτική πολιτική και σε σουηδικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει τίποτα Οι σουηδικέ αρχέ προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα, στράφηκαν και στον ε, Σουηδικό Οργανισμό Περιβάλλοντος με τις ίδιες ερωτήσεις, αλλά ε, πήραν την ίδια απάντηση. Εσείς μας δείξατε έναν κατάλογο με τι, τι χρειάζεται να κάνουν τα κράτη-μέλη για να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο στον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και είναι πάρα πολύ μακροσκελής ο κατάλογος αυτός. Και όποτε κόντευαν να καταφέρουν κάτι στις δικέ αρχές, η Greenpeace έπαιρνε τα πράγματα στα χέρια τη και φτάσανε μέχρι στο να πετάξουν μεγάλες πέτρες, ε, βράχους μέσα στη, στα περιβάλλοντα, στα θαλάσσια, το συγκεκριμένο περιβάλλον. Και μάλιστα δώσανε στις Σουηδικές Αρχές ε, και ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα είχε το να ρίξουν αυτούς τους βράχους ε, στο βοβηθό της θάλασσας. Οι Σουδικές Αρχές δεν έβλεπαν τη δυνατότητα ε, το δικαίωμα να αρνηθούν στην Greenpeace να ρίξει αυτούς τους βράχους. Τώρα ε, ήταν ε, φυσική βράχη ή τσιμεντόληθη. Επειδή δεν ήταν τσιμεντόληθη, αλλά ήταν φυσική βράχη, δεν υπήρχε και κανένας άλλος ε, κίνδυνος. Οπότε η Greenpeace προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή είναι αυτή η οποία ουσιαστικά προστατεύει τις περιοχές Natura 2000 Σουηδία, η Greenpeace. Δεν είναι ιδανική λύση όπως καταλαβαίνετε αυτή. Και γνωρίζω ότι στη Γερμανία το σχέδιο έμπας που αναφέρατε για την υγιή διαχείριση ε, των αλλημάτων στις ε, προστατευόμενες περιοχές έχουν ε, διατρέξει διαξοδικά όλο αυτόν τον κατάλογο Δεν ξέρω ακριβώ τι έχει απαιτήσει από αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως δεν έχουν προτείνει μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε σχόλιο πάνω σε αυτό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε. Γιατί έχει ξεκινήσει όλη αυτή η δυσκίνητη μακροσκελή διαδικασία, αλλά τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Και κάτι ακόμη, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, πραγματικά μας καταθλίβει το γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος μέχρι τώρα δεν έχει εκπονήσει ε, σχέδιο διαχείρισης ε, για το θάλασσο περιβάλλον. Και όταν αφορά τον ειδικό σχεδιασμό για τη θάλασσα, όπως είπατε και εσείς, η Γαλλία δεν εντάσσεται ε, σε αυτά τα σχέδια. Αυτά ήταν τα σχολιά μου. Thanks for that, then, Mrs. Slightly concerned that if... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λόμ. Αν καταστρέφει τα οικοσυστήματα, τα έφραυστα και τα κοράλια αυτή η αλία μετράτες βυθού, ε, τι κάνουν οι πέτρες και οι βράχοι που ρίχνουν μέσα ή που ρίχνει η Greenpeace. Τέλος πάντων, η Greenpeace καμιά φορά έχει περίεργους τρόπους να δραστηριοποιείται. Ο Κρήτον Αρσένης έχει το λόγο. Thank you very much, Mr. Chair. Um, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες φορές και έτσι εντόληθη βοηθάνε. Γιατί σταματούν αυτές τις στράτες. Και δημιουργούν από μόνες τους ένα είδος ε, τεχνητού κοραλιού που βοηθάει να την στο βυθού. Αποφάσισαν τώρα και στην Ελλάδα στα οι κυκλάδες να δημιουργήσουν ε, κάποια πάρκα αλλιευτικά αν θέλετε, δηλαδή κάποιους χώρους ε, προστασίας των αλλιευμάτων, των αλλιευτικών αποθεμάτων. Δεν επιτρέπεται λοιπόν σε προστατευόμενες περιοχές, όπως και σε συγκεκριμένες περιοχές επομένως της Ελλάδας, να ψαρεύει κανείς. Αλλά πριν ε, γίνει αυτή η πρόταση, είχαν δει από τις μελέτες που είχαν να διανεργηθεί ότι η ελευτική δυνατότητα ήταν γύρω από την περιοχή, ήταν τόσο μεγάλη για τους αλείς που τελικά ε, επειδή υπήρχε ελευτική δυνατότητα για τους αλείς, το υποστηρίξανε πάρα πολύ αυτό το, το πρόγραμμα. Δηλαδή η πραγματικότητα για τον Αλιέα θα είναι καλύτερη αν προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές. Προστατεύσουμε και το εισόδημά του. Θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Ποιε είναι οι προθεσμίε για τι χώρε, είπατε για τη Γερμανία ότι θα ξεκινήσει νωρίτερα ε, τον ορισμό των ε, χώρων Natura και μέχρι το 12 θα πρέπει να παρουσιάσουν τα σχέδια διαχείρισης. Ποιες είναι οι κατηγορίες χωρών. Έχουμε αυτούς που ξεκινάνε νωρίτερα ε, και μετά οι υπόλοιποι ξεκινάνε αργότερα. Υπάρχουν τρεις φάσεις. Ε, πώς έχει. Απάντηση. Ουσιαστικά αυτό εξαρτάται από τους ορισμούς των ε, τόπων, των τοποθεσιών. Για αυτούς που θα ορίσουν νωρί, η προετοιμασία πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα σε σχέση με αυτούς που θα πρέπει να ορίσουν αργότερα. Υπάρχει μια εξαετία μετά την έγκριση των προστατευόμενων περιοχών, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για το πώς ακριβώς έχει το διοικητικό υπόβαθρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ωφέλη από τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, αν ήταν αυτή η ερώτησή σας, από το Georgia's Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες ε, ευρείας έκτασης προστατευόμενες περιοχές, γνωρίζουμε ότι η γύρω περιοχή ε, σημείωσε βελτίωση ό,τι αφορά την αλία. Ουσιαστικά επικεντρώνονται οι δραστηριότητες αλίας γύρω-γύρω από την περιοχή αυτή. Βέβαια, ίσως υπάρχουν ε, κάποιες αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία για το περιβάλλον. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι μάλλον πώς, ε, δεν, θα, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι περιοχές, γιατί δεν έχουμε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, δεν έχουμε κάποια διαδικασία μοντελοποίησης για να δούμε τι γίνεται με μικρά τμήματα πληθυσμού σε σχέση με τις μικρές έκτασης αυτές προστατευόμενες περιοχές οι οποίες δεν προστατεύονται κυρίως λόγω των ψαριών, αλλά λόγω τεχνικών εγκαταστάσεων ή άλλων υποδομών που θα πρέπει να προστατευθούν, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάποια πάρκα αιωλικής ε, ενέργειας, αιωλικά πάρκα. Θα πρέπει να οικοτολογήσω για να σας πω ακριβώς. Τώρα, ε, αν θα ωφεληθούν οι αλής Για κάποιες περίκλειστες ζώνες που είχαν οριστεί, παραδείγματος χάρη για, την περιοχή του, για, την, ε, για του Γάδου, έχουμε κάποια στοιχεία. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο για τα πλατήψαρα. Δεν ήταν πολύ σαφέ το αποτέλεσμα ε, για τη, το, στην περίπτωση του Place Box στην Ολλανδία στη Δανία, παραδείγματο χάρη, που δεν επιτρέπει έλλειψη ορισμένων ειδών. Δεν μπορώ λοιπόν να προβώ σε Δεν μπορώ να σα απαντήσω για τι πολύ μικρές αυτές περιοχές, γιατί πολλέ από αυτές τις περιοχές στην Ατούρα 2000 είναι μικρή έκταση. Φαντάζομαι ότι <clears throat> θα υπάρχουν και διαφορές ε, στην Μεσόγειο, όπου έχουμε διάφορα είδη και εκεί θα υπάρχουν διαφορές. Κοιτάξτε, στη Μεσόγειο έχουμε αλληλείς ε, που ζουν εκεί, σε αυτή την περιοχή. Ε, στη Βόρειο Θάλασσα έχουμε όμως ψάρια ε, που μεταναστεύουν άλλα είδη ψαριών και εκεί η κατάσταση βεβαίω είναι διαφορετική. Ως εκ τούτου θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε και διαφορετικά μέτρα. Πρόεδρος, κοιτάξτε, όταν μιλάτε για περιοχές που είναι περίκλειστες, έχουν κλειστεί για προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. <clears throat> Το να αφαιρεί κανείς αυτές τις περιοχές από τους αλείς και ορισμένε είναι πολύ μεγάλες. Έχουν γίνει προσπάθειες αυτές οι περίκλειστες ε, περιοχές ε, να αποκατασταθούν αργότερα. Όταν ε, επισκεφθήκαμε στη Σκοτία τέτοιου είδους περίκλειστες περιοχές. Ήταν κάποιες περιοχές που είχαν σχεδιαστεί για πλατφόρμες εξόριξης. Και είχε όμως σχεδιαστεί και η αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Αυτό εσείς το επιδιώκετε. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλές μελέτες ε, που ασχολούνται με τεχνητούς υφάλους. Ε, ξέρουμε ότι οι πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου προσελκύουν τα ψάρια και επίσης ε, στις περιοχές αυτές αναπτύσσεται και η αλληλεία για λόγους αναψυχής. Όμως για να κάνουμε μια πλήρη ποσοτική αξιολόγηση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για τον Μολύκιο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλακτόν που υπάρχει για την ε, διατροφή αυτών. Όμως ε, για τη Ρέγκα εκεί ε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχει πλανκτό που μεταφέρεται, που μεταναστεύει. Και εκεί είναι μια διαφορετική περίπτωση. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η καταληκτική ημερομιλία για την ολοκλήρωση αυτού του δικτύου του Natura 2000. Τι έγινε, έχει περάσει αυτή η ημερομηνία και διαρωτώ τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν για να διασφαλίσει ότι ε, τα προγράμματα διαχείρισης ε, θα εγκριθούν και θα εφαρμοστούν. Επίσης, διαρωτώ κατά πόσο η Κομισιόν προτίθεται να προτείνει μια πλουστευμένη διαδικασία για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων διαχείρισης. Γιατί αυτή τη στιγμή τα προγράμματα είναι πολύ περίπλοκα και κανένα κράτος μέλος δεν έχει καν παρουσιάσει ένα τέτοιο σχέδιο. Τέλος, ε, διρωτώμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την, ε, ε, τον θαλάσσιο χωροτακτικό ε, σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όπως ακούσαμε στη σημερινή ομιλία και στα συμπεράσματα της παρουσίασης, αυτός ο σχεδιασμός ε, θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της κοινής, μελλοντικής κοινή ελεκτικής πολιτικής. Αυτό είναι και το κλειδί αυτής της ε, πολιτικής. Θα έχουμε μια ολοκληρωμένα θαλάσσια πολιτική, θα προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, θα έχουμε ε, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Αυτά πρέπει να είναι τμήμα ε, μιας μελλοντικής κοινή ελληνικής πολιτικής. Μήπως η Κομισιόν έχει να κάνει κάποια σχόλια επ' αυτού. Έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Γκοντζάλη και τον κύριο Παπούλια. Παπουλία. Ένας από τους δύο ευχαρίστως να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αν ο συνάδελφο ο κ. Παπούλια θέλει να συμπληρώσει, εγώ πάντω θα τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή σε αυτά τα σχόλια. Ε, πάντω θα ήθελα να πω ότι αν θέλει ο συνάδελφο, πολύ ευχαρίστω θα τιμούν ευγνώμων. Λοιπόν, θα ήθελα να, να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση και να πω γιατί τα κράτη-μέλη έχουν τόσο καθυστερήσει όσον αφορά τον ορισμό των σχεδίων ε, ε, διαχείριση για το Natura 2000. Η ερώτηση αυτή ε, είναι πολύ εύστοχη και επίκαιρη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι νοπή συζήτηση ε, πριν από μόλις 10 ημέρες ε, έγινε μια συνεδρίαση με εμπειρογνώμονες Συνεδρίαση ε, ε, ε, θαλασσίων εμπειρογνωμόνων από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλων, οργανώθηκε ακριβώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και κοιτάξτε, πιστεύω ότι το συμπέρασμα αυτή τη συνεδρίαση είναι ότι υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια για να ολοκληρωθεί η διαχείριση αυτή. Κυρίω όσον αφορά τα σχέδια διαχείριση συμπεριλαμβάνοντα με αλληλεπτικά μέτρα. Πρώτον, το πρώτο εμπόδιο είναι Να το πω ως εξή, ότι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Με την έννοια ότι ε, ενώ υπάρχει ε, η πρόθεση από τα κράτη-μέλη να ορίσουν αυτά τα σχέδια διαχείρισης, πολλά κράτη-μέλη περιμένουν να έχουν ένα πιο γενικό πλαίσιο. Δηλαδή, ένα κράτος μέλος αξιολογεί τις απειλές ε, που ε, απορρέουν από την αλία και είναι έτοιμο να προβεί στη λήψη κάποιων μέτρων. Είναι τα προτείνει τα μέτρα αυτά. Έτσι ώστε να εγκριθούν στα πλαίσια της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα φοβάται ότι το γειτονικό κράτος σε αντίστοιχη κατάσταση θα είναι πιο αυστηρό. Μάλιστα πολύ πιο αυστηρό. Και ότι θα πλήττονται τα, τα, τα δικά του τα πλοία τα, και τα σκάφη. Γι' αυτό αμφιβα... διστάζει το κράτο για το κατά πόσο πρέπει να προτείνει τα μέτρα αυτά ή τώρα ή πρέπει να περιμένει η Επιτροπή, μέχρι η Επιτροπή να καθορίσει ένα γενικό πλαίσιο και να οριστούν κριτήρια και μεθοδολογίες έτσι ώστε να είναι σίγουρο τα κρατη για το τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται ε, συναρτήσει των οικοσυστημάτων προς προστασία, των ειδών προς προστασία ε, των ζωνών ε, Natura 2000 πρέπει να προστατευτούν κτλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Η, πρώτη, η απάντηση της Επιτροπής. Τότε, τι να σας πω τώρα. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον και Αλίας, οι δύο γενικές διευθύνσεις, θα, ε, θα, συνεργαστούν για να διοργανώσουν ένα workshop που πρότεινε και η Γαλλία, έτσι ώστε να δαδούν αυτά τα κριτήρια, να συντονίσουν τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζεται κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Και οι επιστημονικοί οργανισμοί και ήδη ο εισηγητή αναφέρθηκε στο ΕΜΠΑΣ και σε άλλα παρόμοια σχέδια. Υπάρχει λοιπόν υλικό αρκετό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε σε κοινοτικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πω καλύτερα, μία κοινή μεθοδολογία. Το δεύτερο πρόβλημα, στο, το οποίο αντιμετωπίζει τα κράτη-μέλη, και αυτό το ανέφερε η κυρία Λόβιν και νομίζω έχει πάρα πολύ δίκιο, είναι λοιπόν η απουσία ενός ε, ε, γρήγορου και αποτελεσματικού μηχανισμού. Ε, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους είχαμε ένα μηχανισμό ο οποίος λειτουργούσε, πώς να το πω, γρήγορα αλλά δεν λειτουργούσε πολύ καλά, έτσι. Όταν ένα κράτος πρότεινε μέτρα, αυτά τα μέτρα προτείνονταν στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο τα ενέκρινε στα πλαίσια του κανονισμού ΤΑΚ, για τα ΤΑΚ, στο παράρτημα 3 με βάση το παράδειγμα 3. Είναι, κάτι που στους νομικούς βέβαια δεν αρέσει ε, ε, ιδιαίτερα, γιατί πρόκειται για διαφορετικά μέτρα από αυτά που θεσπίζονται στον κανονισμό ΤΑΚ. Τέλος πάντων, σήμερα αυτός ο μηχανισμός ήδη δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Επομένως, ο μοναδικός μηχανισμός που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ο, ο συνήθις μηχανισμός στα πλαίσια της κοινή ελευθερικής πολιτικής, που περνά από τη διαδικασία της συναπόφασης και που απαιτεί πολύ χρόνο. Και δεν είναι και αποτελεσματικό. Γιατί, γιατί δεν είναι αποτελεσματικό. Γιατί σήμερα έρχεται η Γερμανία με τι δικέ προτάσει, ένα μήνα αργότερα ή η γαλλια με τι δικέ τη και τελικά δεν μπορούν να εκκρεμούν μία σειρά από διαδικασίε που, είναι, που παίρνουν πολύ χρόνο, είναι χρονοβόρε και περίπλοκε. Η απάντηση λοιπόν και σε αυτό το πρόβλημα ε, είναι κάτι το οποίο επίση αποτελεί αντικείμενο συζήτηση μεταξύ της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, ΜΑΡΕ και Περιβάλλοντος είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ίσως στα πλαίσια της κοινή ελευτικής πολιτικής να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει να αναθέσουμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ανάθεση στην Επιτροπή, ανάθεση στα πλαίσια μιας μελλοντική πιθανής περιφερειοποίησης κοινή ελευτικής πολιτικής, ανάθεση στα κρατημέλη. Όπω ε, έχουν λάβει την εντολή να το κάνουν μέσα στα 12 μίλια. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τι ζώνες, ε, ε τις ζώνε. Και όλα αυτά βεβαίω με τι απαραίτητε εγγύησει. Πώ να το πω, ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με τι επιστημονικέ ενδείξει, με τα κριτήρια, αυτά τα κριτήρια τα οποία αναφέραμε και προηγουμένω κτλ. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν δισταγμού και να μην διστάζουν τα κρατημέλη ω προ την εφαρμογή των, των μηχανισμών αυτών. Τα μελετάμε αυτά και νομίζω ότι θα ολοκληρωθούν ώστε εδώ πιο γρήγορα. Τέλος, θέλω να αναφερθώ το Marine Special Planning στα αγγλικά θα σας το πω, δεν ξέρω πώς το λένε στη γλώσσα μου. Ε, χωροτακτικός θαλάσσιος σχεδιασμός. Ε, η ε, κυρία Λέβιν αναφέρθηκε στο ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα κοινό μηχανισμό για να, για να για να χωρίσουμε σε ζώνες την αλία, στα πλαίσια του συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού. Συμφωνούμε απόλυτα και η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ ακριβώς προ την κατεύθυνση αυτή εργάζεται στα πλαίσια τη ε, ολοκληρωμένη αλληλευτική πολιτική. Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, ένα προβληματισμό για να δούμε πώ όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν αυτό το μηχανισμό. Είναι κάτι το οποίο τολμώ να πω ότι είναι υπερθμόν ένα προτεραιότητα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ε, που μελετάμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος ο Φώτης θέλει να πει κάτι. a few from the να προσθέσω κι εγώ δύο λέξεις από τη ΓΑΜΑ περιβάλλον. Ουσιαστικά την ουσία του θέματος ε, την ανέφερε ο προλαλής σας συναδελφός μου. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να σας καθησυχάσω σε ό,τι αφορά ε, την ε, επέκταση του Natur 2 ε, για τον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι στο επίκεντρο. Είναι μια σημαντική προσπάθεια και για τη διατήρηση της φύσης αλλά και για την επίτευξη των στόχων μας για τη θαλάσσια βιοπικιλότητα. Χαίρομαι επίσης που στο πλαίσιο αυτό έχουμε ολοκληρώσει ένα πλήρες φάσμα θαλάσσιων γεωγραφικών σεμιναρίων. Οι προτάσεις ε, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τα κράτη-μέλη ελέγχθηκαν ε, διεξοδικά σε ό,τι αφορά δηλαδή, τον ορισμό ε, τοποθεσιών περιοχών Natura. Θέλουμε να ξέρουμε και να ξέρουν και τα κράτη-μέλη βέβαια που υπάρχουν προβλήματα για να βελτιώσουν και την έρευνά του τα κράτη-μέλη και να μα δώσουν επαρκή πλήρε προτάσει για την προστασία των θαλάσσιων ειδών και βιοτόπων και οικοσυστημάτων. Τώρα, ταυτόχρονα, αφού είχαμε αυτό το γύρο των γεωγραφικών σεμιναρίων, επικεντρώμαστε και σε ζητήματα διαχείρισης. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος στην πρόσφατη συνεδρίαση με τους εμπειρογνώμονες που είχαμε μαζί με τα κράτη-μέλη, τους εμπλεκόμενους φορείς και από την αλληλευτική κοινότητα και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα δύο αυτά ζητήματα το ένα δηλαδή που έχει να κάνει με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό στο πλαίσιο τη κοινή αλληλευτική πολιτική για την εφαρμογή των μέτρων αλληλεία. Και δεύτερον, μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στι περιοχέ Natura. Όλα αυτά τα είδαμε, τα συζητήσαμε και τώρα συνεργαζόμαστε όλε οι αρμόδιε υπηρεσίε προκειμένου να έχουμε τις ε, οδηγίες που μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη για να τα διευκολύνουμε, όπως βέβαια και στους ε, άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Θα ήθελα να πω ότι τα πορίσματα και οι συστάσεις της έκθεσης αυτής πραγματικά είναι ιδιαίτερως υποδομητικά. θα τα λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη. Τέλος, νομίζω ότι υπήρξε ένα ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρήσουν τα κράτη-μέλη για να ορίσουν ε, τους όρους ε, σύμφωνα με την οδηγία για τους κοτόπους. Ήδη ανέφερε ο συντάκτης της έκθεσης ότι υπάρχει μία περίοδος έξι ετών. Συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα, οι περιοχές ε, ε, στον κατάλογο και μετά έχουν έξι χρόνια τα κράτη-μέλη για να καθορίσουν ε, τα μέτρα διαχείρισης μεταξύ αυτών βέβαια και στον τομέα της αλίας. Δύο στοιχεία όμως που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι πρώτον η πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την εφαρμογή του Natura 2000 που σημαίνει ότι καθυστερεί σημαντικά ε, και η χάραξη των απαραίτητων μέτρων ε, διατήρησης και δεύτερον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να σκέπτονται και να προτείνουν αλλιευτικά μέτρα ήδη από την αρχή. Όταν δηλαδή προτείνουν τους χώρους Natura 2000 για ε, τη θάλασσα συγκεκριμένα, θαλάσσιες περιοχές δηλαδή, να μην περιμένουν να λήξει η εξαετία. Αυτό είναι μια παρότρινση προς τα κρατημέλη και ελπίζουμε να έχει αίσια έκβαση. Okay, thank you very much, uh, Ms. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπούλια και κύριε Γκονζάλης από την Επιτροπή. Ε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και σας κύριε και την ε, παρουσίασή σας και όλους τους άλλους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ίσως λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο σημείο υπαρχμών 14 της ε, ημερήσιας ε, διάταξης. Το 2009 η Ισλανδία ε, μονομερός όρισε μία ποσόστοση για την αλίευση του σκουμπρίου 130.000 τόνων και νομίζω ότι ε, έχει εξαντληθεί πλέον αυτή η, ε, αυτό, αυτό το αλήθεια. Έχουμε λοιπόν τις νήσους ε, Φερόε που παλαιότερα ήταν μέσα στο, εντάσσονταν μέσα στη Συμφωνία για τα Παράκτια Κράτη. Η Ισλανδία βέβαια δεν ήταν γιατί το σκουμπρί δεν υπήρχε στα ύδατα της ε, Ισλανδίας και παραδοσιακά έπαιρναν 2.000 ε, ε, τόνους, φέτος όμως αυξήθηκε σε 130.000 τόνους. Έτσι λοιπόν μετά από διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Νίση Φερόε υπέγραψαν στις 15 Μαρτίου μια συμφωνία που επικυρώθηκε στις 30 Μαρτίου αλλά όμως ε, τελικά οι διαπραγματεύσεις ε, δεν ευβοδόθηκαν, διότι η Ισλανδία και η Νίση Φερό είχαν υπερβολικές ε, απαιτήσει. Λόγω λοιπόν του ότι δεν υπάρχει μία διευθέτηση των ποσοστώσεων ανάμεσα στα παράκτια κράτη, τα επίπεδα αλίευσης αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 900.000 τόνους, είναι πολύ πάνω από αυτό που συστήνουν οι επιστήμονες ως ε, ανώτατο όριο, που είναι 572.000 τόνοι. Γι' αυτό λοιπόν σιγά σιγά φτάνουμε, πλησιάζουμε ε, το 1 εκατομμύριο σκουμπρίου για φέτος Ατλαντικού και αυτό είναι απειλή για το είδος, κάτι που δεν θα ωφελήσει κανένα. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ανησυχίες που εκφράζει ο τομέα τη Αλία ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και γι' αυτό η Κομισιόν ξαναξεκίνησε τι ε, διαπραγματεύσει με την Ισλανδία και τι νήσου Φερόε για αυτό το θέμα. Εγώ πριν από δύο εβδομάδε ε, προσπάθησα να συζητήσω επιτόπου με τι αρχέ των νήσων Φερόε. Επίση μίλησα με τον κύριο Βέσταγκαρτ και με τον κύριο Νίκολσον που ήταν ο πρώην υπουργό. Είχαμε άτυπε συζητήσει για το θέμα αυτό. και οι δύο υπουργοί δέχτηκαν ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτή την περίεργη συμπεριφορά τόσο των Ισών Φερόης όσο και της Ισλανδίας όσον αφορά στα λιεύματα. Και οι δικές μου οι προτάσεις στάλησαν μέσω της κυρίας Φράγκα, της Προέδρου, και στις δύο πλευρές, στους υπουργούς ε, της Ισλανδίας και των νήσων Φερόες, προσκλήθηκαν ε, να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση στις 26 και 27 Οκτωβρίου όταν θα ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό. Στην σημερινή λοιπόν ε, συνάντηση έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Μπάτζινγκ από το Πελασγικό Συμβούλιο και τον εκπρόσωπο των, ε, της Ένωσης Σκοτσέζων Αλλιέων. Ε, η παρουσία επίσης δύο κάμεραμεν οφείλεται στο ότι εκπροσωπούν ε, το BBC Scotland και το STV, ε, τη σκοτσέζικη τηλεόραση. Και βλέπετε λοιπόν αυτό είναι ενδεικτικό για το πόσο πολύ ενδιαφέρεται το κοινό, τουλάχιστον στη Σκοτία. Τα περισσότερα κράτη, παράκτια κράτη που ε, συμμετέχουν σε αυτή την αλία ενδιαφέρονται για το θέμα και αυτό αφορά και πολλά κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν διαφωνείτε λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στους προσκεκλημένους μας και ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βαν Μπάλσφορντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διστάζω να αρχίσω την παρουσίασή μου, γιατί μέρος ε, αυτό που θα ήθελα να πω ε, περιέχεται και στι διαφάνειε. Πάντως πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να αναπτύξουμε κάποιες απόψει εκ μέρους ε, του κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι μέλος του Πελαγικού Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά αυτή τη στιγμή μιλώ εκ μέρους της, του, του Ευρωπαϊκού Πελαγικού, του Ευρωπαϊκού Κλάδου των Πελαγικών Ειδών. Ο τίτλος της μικρής μου παρουσίασης είναι «Διαχείριση του σκουμπριού στο χάο, με χάος, χαοτικό τρόπο», γιατί περί αυτού πρόκειται αυτή τη στιγμή. Πολύ σύντομα να σας πω, εδώ είναι μικρός ο χάρτης, αλλά βλέπετε την κατανομή του είδους ε, στην Βορειοανατολική Ευρώπη και στο δυτικό τμήμα ε, του Ατλαντικού Ωκεανού, ε, στην Βόρεια Αμερική. Αν δείτε όμως λίγο ε, με περισσότερη προσοχή ε, το χάρτη, θα σας πω πώς κινούνται τα αποθέματα. Έχετε το νότιο συστατικό, στον κόλπο, στον πισκαϊκό κόλπο, το δυτικό ε, υποαπόθεμα που, που κινείται πάνω και κάτω στη δυτική ακτή του, της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί αφήνουν τα αυγά τους και μετά πηγαίνουν, μεταναστεύουν στο βορρά και μετά ξαναγυρίζουν ένα μικρό ε, συστατικό βόρεια θάλασσας και μετά έχετε την ε, περιοχή ε, τροφής στο, στο νότιο τμήμα και στη βόρεια θάλασσα και, και στο, βυτικό στο τμήμα. Αυτό επεκτείνεται αυτό το κομμάτι. Και ο χάρτης δεν δείχνει τώρα την Ισλανδία. Δεν υπάρχει λόγος από σύμπτωση έγινε κάτι τέτοιο. Δεν είχε συμπεριλάβει και την Ισλανδία. Τώρα δεν χωράει σε αυτό το χάρτη. Αλλά ο κόκκινος κύκλος, σας πω, ότι περιλαμβάνει και την Ισλανδία. Αν προσέξετε τώρα λίγο περισσότερο το, το σχέδιο διαχείρισης, αυτό υπάρχει εδώ και 11 χρόνια. Και αναδιαρθρώθηκε συνολικά το 2008. Και ε, ε, αυτό εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Έχουμε μια συμφωνία παρακτηων κρατών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Νίση Φερόη από το, από τα μέσα του 90. Και ε, ολόκληρη η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βορρά, Αγγλία, ε, Σκοτία, Ιρλανδία, Δανία, Γερμανία και Νορβηγία, αυτές οι λύσεις και νομίζω και ακόμα και η Σουηδία, όλοι πιστοποιούνται στα πλαίσια των αρχών του MSC από το 2008. Και βεβαίω έχουμε τους ελεγκτές του MSC ε, που ε, ε, μα υποβάλλουν σε έλεγχο ε, σε αιτήσια βάση. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι η διαχείριση του σκουμπριού είναι σχετικά επιτυχημένη. Εδώ βλέπετε τις ε, ε, προσλήψεις ε, στις αρχές του 2000 ήταν μεγάλες ε, και γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το, το απόθεμα είναι μεγάλο. Κοιτάτε τώρα τις εκφορτώσεις. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σταθερές οι εκφορτώσεις. Έχουμε αύξηση τα τελευταία χρόνια, όπω το βλέπετε, και αυτό είναι και μέρο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και, μετά, και τώρα βλέπετε την θνησιμότητα των ψαριών, που αυτή τη στιγμή είναι ε, γύρω στο επίπεδο ε, που θα έπρεπε να φτάσει το 2015 Ήδη το έχουμε φτάσει ε, εδώ και ε, λίγα χρόνια νωρίτερα. Ε, μιλώ με βάση τις αρχές της μέγιστης απόδοσης. Είναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ε, φνησιμότητα. Ε, γίνεται η αναπαραγωγή, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα έλεγα. Τώρα, αν δείτε την ε, βιομάσα αποθεμάτων αναπαραγωγής. Βλέπετε την τάση. Η πράσινη διατηκωμένη γραμμή είναι ε, το επίπεδο στόχου με βάση τη μέγιστη απόδοση, μέγιστη διαρκή απόδοση. Και τα πρόσφατα χρόνια βλέπετε ότι αυτή η βιομάσα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η διαχείριση είναι επιτυχημένη. Αλλά πολύ συχνά στι ιστορίε επιτυχία υπάρχει και ένα αλλά. Και εδώ έχουμε το αλλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Ισλανδία. Η επέκταση των αποθεμάτων έχει να κάνει και με τα περιφερειακά ε, ε, ε, με, με, με, τα περιφερειακά σημεία, εκεί βρίσκεται η Ισλανδία και εκεί λοιπόν επεκτείνεται το σκουμπρί. Και τι έκανε ε, η, Ισλανδία. Άνοιξε την αλία στα, στα ύδατά της, που δεν είναι λάθος από μόνο του. Ελεύθερη λοιπόν αλία μέχρι και το 2009. Και στη συνέχεια, στο υψηλότερο σημείο, 30.000 τόνους, έφεσαν μία ποσόστοση σε αυτό το ακριβώς το επίπεδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για Ολυμπιακό άφλημα, θέλετε. Ε, και αυτό ε, επηρέασε πολύ την κατάσταση. Εδώ λοιπόν ε, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση η Ισλανδία σε σχέση με την ελεύθερη ελεία που ε, είχε μέχρι τότε. Βλέπετε λοιπόν την πολύ απότομη αύξηση μέχρι το 2004 ε, βλέπετε και τα στοιχεία φέτο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια το, έτος, το ελευτικό έτος ακόμα. Πάντως, αυτή είναι μια κατάσταση που θα ήθελα βεβαίω και πολλοί άλλοι να έχουν ε, για τον εαυτό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν. Και το δεύτερο αλλά είναι η νήση Φερόα, που μέχρι το 2009 ήταν εταίροι σε αυτές τις συμφωνίες των παράκτιων κρατών και στη συνέχεια βλέπετε το μερίδιο που είχαν, ε, το ποσοστό, το, το 4,6% του συνολικού ΤΑΚ, που φέτος είναι 26.000 τόνοι. Ε, μπορεί να λείπουν λίγοι τόνοι εδώ, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι το... για αυτή την τάξη μεγέθους. Και στη συνέχεια έφυγαν από τη Συμφωνία των Παράκτιων Κρατών 2010. επειδή υπήρχε ένα αίτημα για, για υψηλότερο μερίδιο μέχρι το 10%. Αλλά δεν συμφωνήθηκε με του εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νορβηγία. Έφυγαν λοιπόν από αυτή τη συμφωνία. Και, για να μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ισλανδία, όσον αφορά την ελεία του, του σκόμβρου. Πριν, λίγες μέρες λοιπόν πριν τις διακοπές έθεσαν με ποσόστοση 85.000 τόνων που είναι ε, τρεις φορές το κανονικό μερίδιο. Και μετά έχουμε μια μεγάλη χώρα, αλλά ως προς το σκουμπρί μικρή θα έλεγα. Είδε την κατάσταση αυτή και τις εξελίξεις αυτές η Ρωσία. Και εκεί, επειδή η συμφωνία για το σκουμπρί κατέληξε σε μια συμφωνία και είχε πολύ μικρό ε, ποσοστό, και έθεσε τώρα ένα αυτόνομο ποσοστό που είναι το διπλάσιο περίπου από το κανονικό μερίδιο. Άρα και η Ρωσία ακολούθησε αυτήν την τακτική. Οι επιπτώσεις όλων αυτών είναι ότι θα μπορούσαν να είναι καταστροφικέ θα έλεγα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. όπω είπα και πριν από λίγο, η θνησιμότητα των ψαριών δεν παρουσιάζει πρόβλημα μέχρι φέτο. Παρά το γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν προσορίσει σε επιπλέον αλλιεύματα, δεν χτύπησε κόκκινο η θνησιμότητα των ψαριών. Τα πράγματα εξακολουθούν ακόμα να είναι εντάξει. Γιατί όπως σας είπα, επεκτείνονται τα, τα αποθέματα, έχουμε καλούς, καλά ποσοστά αναπαραγωγής και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δείτε τώρα τι γίνεται το 2010, η, συμβουλή, η επίσημη συμβουλή ήταν ΤΑΚ ήταν 572.000 τόνου. που δεν ε, είναι μικρότερο από το 2009. Το απόθεμα αυξανόταν, αλλά ε, η συμβουλή ήταν να πάμε για χαμηλότερα ποσοστά. Γιατί ο βασικός λόγος είναι ότι τα αλλιεύματα θα είναι ψηλότερα από τα προβλεπόμενα από την επιστημονική κοινότητα λόγω των αυτόνομων ποσοστώσεων που έθεσαν η Ισλανδία, για παράδειγμα. Και οι νήσοι Αν τώρα δείτε την κατάσταση του 2010, δεν έχουμε πλέον παράκτια συμφωνία, γιατί έφυγαν και οι νήσοι και η Ισλανδία δεν ήταν μέρος έτσι κι αλλιώς. Άρα στην τελευταία ανάλυση μπορούμε να μιλήσουμε, και αυτό έγινε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία κινήθηκαν προς μια διμερή συμφωνία που συνήφθηκε νομίζω το Φεβρουάριο αυτού του έτους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία ακολούθησαν την, ε, συμβουλή, την επιστημονική συμβουλή και ε, πήραν το κανονικό μερίδιο των, των προηγούμενων χρόνων, 572.000 τόνοι, ε, που ήταν η συμβουλή του ISIS. Επίσης το ISIS υπολογίζει ότι φέτος το συνολικό αλλιεύουμε στην τελευταία ανάλυση, γιατί προβλέψουν όλα αυτά, έτσι, ότι θα είναι γύρω στις 930.000 τόνους, που είναι 60% περισσότερο από ότι η, η συμβουλή που ε, έδωσε το ΙΣΕΣ και που έγινε και, και δεκτή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νορβηγία. Επίσης, 2010 έχουμε ε, την, αυτή την ε, πολύ δαπανηρή έρευνα για τα αυγά. Βρίσκουμε την παραγωγή αυγών και με βάση αυτή την παραγωγή αυγών έχουμε ένα πολύ καλό δίκτυο για το μέγεθος των αποθεμάτων. Το αποτέλεσμα αυτής της ε, έρευνας δείχνει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το απόθεμα. Το 2007 έχει γίνει τελευταία έρευνα αυγών. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα ε, της ε, συμβουλής του ΆΙΣΕΣ. Να δούμε πόσο αυξήθηκε, αλλά υπολογίζουμε γύρω στο 20%. Αλλά εάν προσέξει κάπως καλύτερα τα στοιχεία, θα δει ότι η παραγωγή αυγών στην Κοιτάξτε, ε, η παραγωγή των αυγών γίνεται ακριβώς εκεί όπου αφήνει τα αυγά του ε, το ψάρι. Και βλέπουμε ότι η παραγωγή αυγών στην Ισλανδία ε, είναι το 0,3% του συνολικού. Και η παραγωγή αυγών στις Φερόες είναι το 0,7% του συνολικού. Πολύ μικρό ποσοστό και εδώ. Μόλις 0,7%. Βλέπετε λοιπόν, και θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η αναπαραγωγή του σκουμπριού γίνεται, και αυτό είναι σαφές, στα ε, ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 99%. Και εδώ βλέπετε, είναι μικρές αυτές οι εικόνες, αλλά και τα αυγά είναι μικρά, έτσι. Και βλέπετε εδώ ε, ότι ε, που, που έχουμε την κατανομή των μεγάλων ζωνών αναπαραγωγής. κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης η οικονομική ζώνη στις νήσους Φερόας και στο κίτρινο είναι ε, ε, η ζώνη της Ισλανδίας. Και βλέπετε πότε έγινε η έρευνα, τότε που είναι ορατά τα αυγά. Αυτό είναι η απόδειξη. Ότι δηλαδή ε, οι ζώνες αναπαραγωγής γίνονται, είναι, είναι βασικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν στην Νορβηγία. Not only this year, but last year and all... Ε, ακόμα και πριν τρία χρόνια, είχαμε ε, αναρωτηθεί για το τι γίνεται και στις, ε, στις νήσους Φερός και στα, στην Ισλανδία. Γράψαμε λοιπόν μία επιστολή προς, τον, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ληφθεί συγκεκριμένη δράση κατά της Ισλανδίας και των νήσων Φερός. Βεβαίω, ω βιομηχανία είμαστε ελεύθεροι να, υποβάλουμε, να ζητάμε ό,τι θέλουμε. Αυτό που ζητούσαμε και να υποβάλουμε έτοιμα για ό,τι θέλουμε ήταν, να, ζητούσαμε από τότε να σταματήσει αμέσως η διμερή συμφωνία με τις νήσους Δηλαδή, καμία ε, πρόσβαση ε, πέραν των χιλίων τόνων, που ήταν μέρος της ε, συμφωνίας. Και θα έπρεπε πρώτα... Και, και κοιτάξτε, σε ορισμένες περιόδους του χρόνου μπορεί να γίνει ελεία μέχρι το Φεβρουάριο και από τον Οκτώβριο και μετά. Ίσως λοιπόν έχουν, έχουν ακόμα έχουν ε, μέχρι στιγμής ψαρέψει 85.000 και ε, απομένει ακόμα και ένα μεγάλο μέρος βάσει της ημερούς ε, συμφωνίας. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά είναι κάπως παράδοξο. Ε, Γι' αυτό ζητάμε να ανασταλεί αμέσω αυτό το τμήμα τη συμφωνία και να ληφθούν ε, κυρώσει. Θέλουμε να κλείσουν τα λιμάνια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ζώνε, ε, να κλείσουν σε όλα τα ε, ε σκάφη τη Ισλανδία και, ε, και των ίσων Φερόε να ε, μπουν σε ένα μαύρο κατάλογο, στο μαύρο κατάλογο της ε, παράνομη και άναρχης ε, να υπάρξει άμεση αναστολή από, από την Ισλανδία ε, το, της δηλωμένης ποσόστοσης κόμβρου των 130.000 τόνων, ε, έτσι όπως προβλέπεται στις ε, ε, διαπραγματεύσεις ένταξης που ξεκινούν σήμερα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έγινε τίποτα. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι η οικονομική άποψη είναι όλα αυτά αδύνατα από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι ξέρουμε δεν έχει λεφθεί καθόλου καμία δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι ξέρουμε, έτσι το τονίζω. Τελειώνω λοιπόν την ομιλία μου λέγοντάς σας ότι ότι δεν γίνεται σχεδόν καθόλου αναπαραγωγή στα, ε, στη ζώνη αυτή, τη, στη ζώνη αλίας της Ισλανδίας και των Ίσων Φερόες. Ε, ο μόνος λόγος τον οποίο ε, η αλία στην περιοχή αυτή είναι επειδή ε, επεκτείνεται για να πτήσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα το απόσταμα και μετακινείται και στα ύδατα αυτά. Και βεβαίως, επίσης πιστεύουμε ότι, και συμφωνούμε ότι η Ισλανδία έχει το δικαίωμα να είναι παράκτιο κράτος βεβαίως. Και ναι, πρέπει να πάρει ένα κάποιο μερίδιο, ένα κάποιο ποσοστό του ΤΑΚ, αλλά, και αυτό για μας είναι το βασικό σημείο, δεν θα πρέπει να δίδεται πρόσβαση στην Ισλανδία στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά πιστεύουμε, το είδαμε και με το προσφυγάκι, αν είναι ε, πολύ γρήγορο, ε, κυρίως ε, τα, τα, τα, τα ενδυμικά είδη, όπως το σκουμπρί, τα οποία κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, ψάχνουν διατροφή και ε, μετακινείται προς τα έξω, ενώ όταν συρρυκνώνεται ξαναγυρίζει πίσω. Αν δώσουμε λοιπόν πρόσβαση στην Ισλανδία για το δικό του το μερίδιο του, του σκόμβρου, τότε ακόμα και όταν έχει μειωθεί ε, ε, ε, το απόθεμα και έχει φύγει από τα ύδατα, θα εξακολουθήσουν το ψαρεύουν στα δικά μας τα νησιά. Το είδαμε αυτό να γίνεται και με το προσφυγάκι. Γιατί η Νορβηγία, για παράδειγμα, είχε μεγάλο μερίδιο του, του ΤΑΚ για το, ε, για το, για το είδος αυτό. και στη συνέχεια, όταν μειώθηκε, άρχισαν να έρχονται στην Ιρλανδία. Αυτή τη στιγμή θέλουμε μια προσωρινή συμφωνία, γιατί το απόθεμα κινείται ιδιαίτερα. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται. Και δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε αν αλλάξουν ε, τα πράγματα σε τρία χρόνια, όταν θα γίνει η επόμενη έρευνα. Και αυτό είναι θέμα τακτικής βέβαια περισσότερο. Τώρα έχουμε μια συμφωνία ε, για το σκουμπρί δεκαετή με την Ορβηγία. Και όλοι όσοι συμμετείχαν στι διαπραγματεύσει με την Ισλανδία και τι νήσου Φερόες, του καλώ να συνεργαστούν με την νορβηγική κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, τα, τα συμφέροντά μα είναι τα ίδια με τα συμφέροντα τη Νορβηγία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τα ίδια. Άρα μα συμφέρει να συνεργαστούμε ιδιαίτερα στενά με την Νορβηγία. Και εμεί, ω κλάδο, συνεργαζόμαστε ιδιαίτερα με τον αντίστοιχο κλάδο τη Νορβηγία. Και αυτό είναι συμβολική σημασία βέβαια, δεν είναι πολύ σημαντικό. Σα παρακαλούμε μην αφήσετε, βγάλτε ε, τη δυνατότητα να έρχεται και να, λιεύει, ε, να λιεύουν οι νήσοι Φερόε στα, ε, στα ύδατά μας. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους Να τους αφήνουμε δηλαδή, όταν πήραν το τριπλάσιο, να, να, να, να μην του αφήσουμε πλέον από τον Οκτώβριο και μετά να ψαρέψουν τίποτα. Και σα παρακαλώ, μην ξαναγίνει η ιστορία αυτή η δραματική κατάσταση που έγινε και με το προσφυγάκι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. That's quite presentation. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Σκοτσέζικης Οργάνωση. Ian Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολή γιατί μπορεί να επαναλάβω κάποια από όσα είπε ο συνάδελφο. Ίσως όμω να χρειάζεται και να τα επαναλάβω. Το απόθεμα σκουμπρίου είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και γιατί έχει κάποιες οικονομικές πτυχές, γιατί έχει κάποιες πτυχές που σχετίζονται με τη διαχείριση. Είναι ίσως το πιο εύθραυστο, το πιο τροτό Το 2010 είχαμε γύρω στους 367.000 τόνους για να αλλιεύσουμε και η μέση τιμή για, τον, για την πρώτη πώληση ήταν 10.000 ευρώ. Άρα μπορείτε να εκτιμήσετε πόση αξία είχε το 2010. Ήταν γύρω στα 370 εκατομμύρια ευρώ για το 2010 η αλία του σκουμπριού. Η Ολλανδία έχει 29, η Δανία, η Ισπανία είχαν 29, 28 μάλλον εκατομμύρια, με 14 συνολικά κράτη-μέλη να έχουν δικαίωμα αλήψης των αποθεμάτων του σκουμπρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, θα πρέπει να θεωρηθεί πραγματικά το κόσμημα της αληφτικής διαχείρισης, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα. Πραγματικά πάνω από 20 χρόνια έχουμε πολύ επιτυχή διαχείριση των αποθεμάτων και έτσι μπόρεσε το απόθεμα να επεκταθεί και να αναπτυχθεί και βορειοδυτικά μεταξύ της ε, Σκοτίας και των Φερόε στην, ε, και στην ε, θερινή περίοδο. Βέβαια υπάρχει η μετακίνηση του αποθέματος προς τα βορειοδυτικά λόγω της θέρμανσης του πλανήτη αλλά υπάρχει και το εξής. Εάν υπάρξει προσεκτική ασφαλής ε, μακροδιαχείριση, τότε θα μπορεί να γίνει ασφαλής μετακίνηση του αποθέματος. Θεωρούν ε, τα Φερόε και η Ισλανδία ότι κάνουν ε, καλή διαχείριση. Επιτρέπουν όμως την αλίευση των αποθεμάτων όταν είναι στα ύδατά τους χωρίς κανένα περιορισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 367.000 ε, τόνους ποσόστοση, όπως είπα. Αν όμως μπορεί ο αλλιευτικός μας στόλος να ψαρεύει όπως ο Ισλανδικός, μπορεί να φτάσει να αλλιεύει εύκολα και ένα εκατομμύριο σκουμπρία. Είμαστε υπεύθυνοι όμως και δεν το κάνουμε αυτό, γιατί θέλουμε τη βιώσιμη αλία. Θέλουμε να παραμείνει το απόθεμα, να είναι βιώσιμη η αλληλεία και να την περάσουμε και στην επόμενη γενιά των Σκοτσέζων αλλιέων αυτή τη δραστηριότητα. Τι κάνουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια. Οι μακροελιό, όπως είπε και ο συνάδελφος, ε, πραγματικά μπορούν να ε, επαληθευθούν και έχουν επαληθευθεί ε, ότι είναι και παραδείγματα καλής διαχείρισης και παραδείγματα βιωσιμότητας. Η ανεύθυνη όμως δράση των Φερόε και της Ισλανδίας δημιουργεί προβλήματα. Πραγματικά ο ιστός, ο κοινωνικός των αλλιέων κινδυνεύει στη Σκοντία και θέλουμε να κληρωθούν τα αιτήματα των αλλιέων. Έχουμε πολλά, πολλές συνιστώσεις. Έχουμε τους αλλιείς οι οποίοι ψαρεύουν πάνε στη θάλασσα. Χρειαζόμαστε καλούς αλλιείς, χρειαζόμαστε επίσης και την διατήρηση των αποθεμάτων επιτόπου, ναυπηγεία, ηλεκτρισμός. Πάρα πολλοί κλάδοι ζουν από τη δραστηριότητα αυτή και φυσικά και πρέπει να έχουμε και μια πάρα πολύ καλή και ε, ανθούσα μεταποιητική βιομηχανία. Όλοι αυτοί οι κλάδοι λοιπόν ε, εξασφαλίζουν ε, θέσεις απασχόλησης για την κοινότητα. Αλλά το σημαντικότερο θέμα που είναι πάνω απ' όλα είναι το δικαίωμα των αλλιών. Αν δεν έχεις ποσόστοση, πώς να έχεις και μια επιτυχημένη αλλιευτική κοινότητα. Σκοτία πολλοί έχουν χάσει το εισόδημά τους και πολύ ίσως να θυμόσαστε ότι είχαμε με την Ισλανδία ένα είδος ε, ψυχρού πολέμου, ε, μάλλον είχαμε ένα είδος πολέμου με τον, για το γάδο. Ε, και ξέρουμε πόσο μεγάλη αλληλευτική δραστηριότητα γίνεται στα Ισλανδικά ύδατα. Οι αλληλείς που παλιά είχαν πάρα πολύ ανθυρή οικονομική κατάσταση είναι η σκιά του εαυτού τους πλέον και η μεταπητική βιομηχανία πραγματικά έχει οδηγήσει σε κατάρρευση την αλληλευτική κοινότητα και έχουν χάσει πραγματικά τις αλληλευτικές τους, τα αλληλευτικά τους δικαιώματα. Εξ αυτού, επ' αυτού πρόκειται λοιπόν, πρόκειται για την επιβίωση της αλληλευτικής κοινότητας της Σκοτίας και το ίδιο ισχύει και για πελαγικά λιμάνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Ελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της τη διαφορά που έχουμε και χαιρόμαστε και πραγματικά είμαστε γνώμονες στην Επιτροπή σας που κάνετε ό,τι μπορείτε για να προστατεύσετε το πολύτιμο αυτό απόθεμα και όλα όσα διακυβεύονται. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε πραγματικά να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει συμφωνία, γιατί σίγουρα είναι προ όφελο όλων, αλλά αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί περισσότερο είναι ότι η κληρονομιά των αλληλευτικών μα δικαιωμάτων να μην δοθεί αλλού. Πολύ απλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. You made a very important and pertinent... Πραγματικά ήταν πολύ εύστοχα και πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Πράγματι μιλάμε για ε, πολύ καλή διαχείριση και ίσως είστε μια μοναδική περίπτωση που έχετε ακριβώς αυτή την πιστοποίηση του MSC ότι κάνετε καλή διαχείριση. Δηλαδή το 80% των αποθεμάτων να χαρακτηρίζονται από η επεραλίευση, εσείς έχετε καταφέρει ε, βιώσιμη αλυσία που πιστοποιείται και από το ΕΜΣΥ. E Λόγω των προσπαθειών ακριβώς ε, των ε, Ευρωπαίων αλιέων στην πελαγική αλία και φυσικά και των Ορβηγών αλιέων που πραγματικά έχουν πληρώσει σε ό,τι αφορά και την καλή διατήρηση μειώνουν τις ημέρες ε, κατά τις οποίες ε, βγαίνουν ε, στα νερά, στα ύδατα για να ψαρέψουν, σέβονται τις επιστημονικές συμβουλές, μειώνουν τις ποσοστώσεις τους. Και τώρα έχουμε τα Φερόε και την Ισλανδία να κάνουν ό,τι θέλουν, ουσιαστικά καταστρέφοντας τις δικές μας προσπάθειες διατήρησης των αποθεμάτων. Και δεν με εκπλήσει σε καμία περίπτωση το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση και πολύ μεγάλη αγανάκτηση και θυμός. Είχαμε πριν από κάποιες εβδομάδες εδώ και ένα είδος ε, του αποκλεισμού ενός ε, σκάφους ε, ε, πελαγικού από τα Φερόε. Δεν μπόρεσε να εκφορτώσει, το απέτρεψαν οι αλλοί τη περιοχή. και μετά από διάφορες, από αρκετές ημέρες ε, που αφήγε καταστραφεί ως φρέσκο, ως νοπόψάρι το απόθεμα, το, θα, μπορούσε μόνο να το χρησιμοποιήσει για ηχθιάλευρα. Και η κυρία Δαμανάκη, Επίτροπος, είπε ότι κατάλαβε την αυθόρμητη αυτή αντίδραση των αλλίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πραγματικά παλεύουν για τη ζωή τους, για την επιβίωσή τους, για το εισόδημά τους. Όταν ε, μίλησα στους υπουργού πριν από κάποιες εβδομάδες με τους Υπουργού των Φερό και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα συνάντησα και τον ε, Ισλανδό πρέσβη, στο Στρασβούργο ε, μου είπαν στα Φερόε ότι έχουν ε, πάρα πολύ μεγάλα ε, αποθέματα γάδου και βακαλάου, αλλά η μεγάλη, η μαζική ποσότητα των σκουμπριών ουσιαστικά επιτίθενται και τρώνε τους νεαρούς γάδους. Και γι' αυτό δεν έχουν μεγάλο απόθεμα σε σκουμπρί. Τέλο πάντων αυτό έλεγαν και γι' αυτό είπαν ότι πρέπει να ε, ψαρεύουν ε, τον, ε, το σκουμπρί για να μην τρώει τα άλλα Και ο Ισλανδός πρέσβης μου είπε ότι στην Νότια Ισλανδία υπάρχει και, άλλη, και άλλο ένα είδος το οποίο μειώνεται Πάφιν είναι η αγγλική του ονομασία. Λόγω των αμόχελων, που είναι και η βασική τροφή τους και τα οποία δυστυχώς μειώνονται. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα και τα νησιά Φερόε και η Ισλανδία πάντοτε περηφανεύονται για την αλία τους και πόσο καλά τη διαχειρίζονται και πόσο βιώσιμη είναι. Να ε, λειτουργούν όμως τόσο αυθαίρετα και να ορίζουν τις μονομερείς αυτές ποσοστώσεις είναι πραγματικά κάτι απαράδεκτο. Νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική συμφωνία. Πρέπει, και συμφωνώ με τους δύο μιλητές, πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Δεν μπορεί να συγχεχιστεί και να έχουμε τα ίδια πράγματα και του χρόνου. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι τελικά επιβραβεύουμε κακές πρακτικές. Δεν μπορούμε να πούμε απλά στην Ισλανδία και στα Φερόε. Ωραία, μάλιστα αυξήσατε με αυθαίρετο τρόπο τις ποσοστώσεις ε, σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα και θα σας δώσουμε αυξημένες ποσοστώσεις σε επόμενες ε, συμφωνίες με παράκτη κράτη και θα δώσουμε τελικά σε αυτές τις δύο χώρες πρόσβαση στα νέα υδατά μας και πάλι. Αυτό είναι απαράδεκτο να το κάνουμε. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι τα νησιά Φερόε δεν είναι και πολύ ικανοποιημένα με αυτή την κατάσταση, ότι είναι εκτός δηλαδή της συμφωνίας με τα παράκτια κράτη και ίσως, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, ίσως επιτελέσουμε κάποια πρόοδο ε, ίσως καταφέρουμε να τους προσκαλέσουμε ξανά σε αυτή τη συμφωνία. Και σε ό,τι αφορά αυτή την τριετή έρευνα για τα αυγά, που δείχνει σημαντική αύξηση των αποθεμάτων, ίσως η ISIS κάνει κάποιες διαφορετικές προτάσεις για τα νησιά φερογιά του χρόνου. Και ούτω ή άλλω, όπως έχουν οι ποσοστώσει του τώρα μπορεί να πάρουν ε, μια αύξηση αν ε, για το χρόνο. Τώρα η πρόσβαση τη Ισλανδία στα δικά μας ύδατα αυτό είναι απαράδεκτο και αποκλείεται να γίνει. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε σε καμία περίπτωση υπό κανέναν όρο για όλου αυτού του λόγου ο οποίο ανέφερε ο κύριος Μπάλφορ. Ούτε ήξερα μέχρι να μου το πείτε το μεσημέρι στο γεύμα και το είπατε και επανειλημμένο στην παρουσίασή σας. Ούτε και ήξερα λοιπόν ότι η συμφωνία προβλέπει ότι θα πρέπει να δίνουμε 4.600 460 συγγνώμη, χιλιάδες τόνους By the fact... 4.600 τόνους μια τους ψαρεύω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε αυτό. Το είπα στον ε, κύριο Φαμπάλσφορ όταν μου το είπε το μεσημέρι. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε, μας κλέβουν μας, ε, οι διαρρήκτες στο σπίτι μας και την ώρα που φεύγουν τρέχουμε για να τους δώσουμε και αυτά που ξεχάσανε. Πώς μπορεί η Κομισιόν να πει στα Φερόε Συγγνώμη, δεν θα πάρετε 4.600 επιπλέον τόνους, δεν το αξίζει η συμπεριφορά σας. Γιατί να μπορεί να το πει αυτό. Λοιπόν, πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Κτιμώ ε, την κατάσταση. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κ. Σπένσερ και η Επιτροπή. Σίγουρα μπροστά και πισωρέμα για αυτούς. Αλλά πρέπει να καταλήξουμε στην τριμερή συμφωνία με Φέρο Νορβηγία Ευρωπαϊκή Ένωση, απομονώνοντα την Ισλανδία, εάν δεν είναι προετοιμασμένοι να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κατά προτίμηση, θα ε, θέλαμε μια τετραμερή συμφωνία. Όχι όμως να επιβραβεύσουν ουσιαστικά την κακή συμπεριφορά χωρίς να είμαστε σκληροί στην αντιμετώπιση μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και επίσης ευχαριστώ και τους ε, προσκεκλημένους μας ε, για τις ε, πολύ περιεκτικές και κολονόητες για μένα τουλάχιστον παρουσιάσεις. Δεν θέλω να παραλάβω αυτά που λέχθησαν. απλά θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε αυτό που θα μπορούσε ή αυτά που θα μπορούσαν να είναι περισσότερο πολιτικής χρειάς θέματα. Ε, βλέπω ότι πολλοί ε, πλέον έχουν κοραστεί με αυτή την μόνιμη δίθεν ε, δυναμική και άποψη ότι εμείς οι Ευρωπαίοι συμπεριφερόμαστε σωστά και άλλοι λάθος. Έχουμε εμείς καθορίζουμε τα λεύματα και άλλοι τα καταστρέφουν. Έχει φτάσει λοιπόν νομίζω η στιγμή να δούμε τι θα ήτανε πιο σκόπιμο και ποιο θα ήταν το καλύτερο απόθεμα να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό και νομίζω ότι έχει φτάσει στιγμή να τοποθετηθεί και η Κομισιόν. Ακούσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαν να κλείσουν ε, τα λιμάνια για τις εκφορτώσεις ε, από την Ισλανδία. Βεβαίως και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει η Κομισιόν. Αν η Κομισιόν επιθυμεί να περιμένει τη νομική ασφάλεια ε, να αποφασίσουν τα δικαστήρια. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα συνεχιστεί η κατάσταση, θα υπάρχει ε, λαιλασία αυτών των ε, ε και η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά. Θέλω να το πω αυτό για την ε, κοινιαλευτική πολιτική. Παρότι σε αυτή τη συνάντηση δεν μιλάμε τόσο για την κοινιαλευτική πολιτική, όμως η αξιοπιστία της εξαρτάται από τις ε, ενέργειες ε, που λαμβάνει η Κομισιόν. Αν η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα, τότε το σύνολο της αλληλευτικής πολιτικής δυσφημείται όλο και περισσότερο. Γίνεται αναξιόπιστη αυτή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη φάση και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μια νέα πολιτική. Αν λοιπόν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, ε, οι άνθρωποι, ε, οι υπόλοιποι απλά θα ε, γελούν εις βάρος μας. Όσον αφορά την οξιοπιστία μας, εχθές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μιλήσαμε λιγάκι για το θέμα αυτό, ρωτήσαμε την Επίτροπο και εκείνη είπε ότι δεν βλέπει πώς οι συζητήσεις για την ένταξη της Ισλανδίας θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτό ή αυτό το θέμα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Όμως, εφόσον το, η αξιοπιστία είναι ένα κρίσιμο θέμα, γιατί όχι. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω από την Κομισιόν κατά πόσον την επόμενη εβδομάδα που θα πάει στην Ισλανδία για ενταξιακή επίσκεψη, κατά πόσον έχει συμπεριλάβει το θέμα και αν όχι, γιατί όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τις ε, πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για αυτή την τραγική κατάσταση, πρέπει να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να εκτελείστε μία τραγωδία. Μάλιστα θα έλεγα ότι είναι μία κλασική περίπτωση για το πώς ε, κακοδιαχειριζόμαστε τα ληφτικά αποθέματα ανά τον κόσμο. Κυρίως όμως αυτά που μεταναστεύουν όπως είναι ο ε, ο τόνος, ε, ε, τα ψάρια αυτά αφήνουν τα αυγά τους σε μία περιοχή και μετά μεταναστεύουν. Είναι λοιπόν δύσκολο για ένα κρατος μέλος να ορίσει ακριβώς το ποια θα πρέπει να είναι η ελευτική δραστηριότητα. Τα ψάρια λοιπόν μεταναστεύουν. Στο τέλος η ελήψη γίνεται από ένα άλλο κράτος μέλος. Όσο λοιπόν υπάρχουν ψάρια στη θάλασσα, αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Και θεωρώ ότι εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου μια ευρύτερη εικόνα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Να ενισχύσουμε τις αλληλευτικές κοινότητες και να δούμε λιγάκι και την διεθνή διαχείριση των αποθεμάτων, όπου υπάρχει κοινή διαχείριση. Γιατί και αν ακόμα ε, μπει η Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ίσως την υπόθεση την κερδίσουν οι νήσοι Φερόες. Και ό,τι και να γίνει θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για την τελευταία φορά. Αυτό το πρόβλημα αφορά πολλά αποθέματα και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ένα πολύ καλύτερο σύστημα κυρώσεων σε διεθνές επίπεδο και να έχουμε και καλύτερα εργαλεία διαχείρισης. Ο κύριος Στίβενσον μας μίλησε για την Ισλανδική εκδοχή ε, των γεγονότων ε, για το σκουμπρί, για τους ε, νεογνούς γάδου. Αυτά όμως είναι παράδειγμα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οικοσύστημα με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Έχουμε ακούσει και κατά το παρελθόν τα ίδια επιχειρήματα από την Ισλανδία για τις ε, φάλαινες, ότι οι φάλαινες ε, τρώνε το γάδο, ότι ε, υπάρχει εκεί απειλή κατά της φάλαινας και πολλά παρεμφερή. Αυτά λοιπόν τελικά καταλήγουν ότι αν δούμε λιγάκι την προσέγγιση για το οικοσύστημα, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ωκεανούς, με μεγάλες θαλάσσιες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να παραμένει ε, άκαμπτη στη θέση της, να ενισχύσει και τις αλληλευτικές κοινότητες και την διαχείριση των αποθεμάτων. Και θέλω να αναφέρω και άλλα δύο θέματα. Ίσως ε, να έχουμε σε ευρωπαϊκά ήρετα τοκια σκουμπριού. Αλλά δεν ισχύει αυτό για όλα τα είδη. Πολλά ε, ε αφήνουν τα ψάρια τους σε, σε που είναι πολύ, πιο μακριά, πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή το επιχείρημα αυτό δεν ισχύει για όλα τα ψάρια. Ας πούμε η περίπτωση του γάδου και εκεί είναι τελείως διαφορετική η οτοκία. Και κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μια συζήτηση με κάποιον από τις νήσιους Φερόες, γιατί δεν μπορούμε απλά να εικάζουμε ποια θα ήταν η απάντησή τους. Πρέπει να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση με τους ίδιους για το θέμα αυτό. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την ευρωπαϊκή εκδοχή των γεγονότων, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο επιδημητικό ε, να ακούσουμε από τους ε, ίδιους την άποψή τους. Προτείνω η Κάρμεν Φράγκα να προσκαλέσει ε, τον Υπουργό Αλίας και τον Υπουργό Εξωτερικών και των δύο αυτών περιοχών στην επόμενη συνεδρίαση. Ε, κοιτάξτε, ήδη έχουν σταλεί προσκλήσει, αλλά δεν προλάβα να έρθουν σήμερα. Πάντως έχουμε προσκαλέσει στις 27 Οκτωβρίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψή του. Ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε κάποιες θετικέ εξελίξεις, γιατί στις 20 ε, Οκτωβρίου ε, θα γίνει μια πολύ μεγάλη σημαντική συνάντηση ε, σε επίσημο επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο και ελπίζω να έχει υπάρξει πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, ε, ε, πιστεύω ότι ήταν καλό να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων με του ενδιαφερόμενου υπουργού. Και βεβαίω, αν συμφωνήσουν και ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μα, θα έρθει. Θα έρθουν. Ο Μισελ Καντέκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ του ομιλητέ που μα ξεκαθάρισαν το θέμα. Νομίζω ότι σχεδόν όλα ελέγχθησαν Προσπάθησε ο προσεκλημένος μου να μας εξηγήσει την κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια ε, καταβάλει έννοιες προσπάθειες για την προστασία των ειδών και καλά κάνει, αυτό θα κάνει και στο μέλλον. Νομίζω ότι αν δεχθούμε αυτό το, ε, ε, αυτό το πραξικόπημα από τις, κατά κάποιο τρόπο από ε, τις και την Ισλανδία, θα βλάψουμε ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή πολιτική. Από την άλλη μεριά, όπως είπε ο συνάδελφος Γκέρινγκ και εδώ, ε, σας το λέω και υπενθυμίζω, ότι είναι υποψήφια η προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τέτοια στάση ε, νομίζει ότι θα διευκολύνει την ε, είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τις υποστηρίξουμε. Άλλωστε αυτή η στάση, αυτή η επίδειξη ισχύω δεν της δίνει ατού και πλεονεκτήματα για την ένταξή της. Νομίζω ότι και όσου προσδοτήτη με αυτό και ω προ άλλα, δεν πρέπει να μας τα λόγια μα. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, σαφεί, αποφασιστικοί και να μην δεχθούμε που δεν είναι λόγο τέτοιε συμπεριφορέ ε, ε, από ε, τι χώρε αυτέ. Είναι παράδεκτο. Όσον αφορά το σκουμπρί που τρώει τα, τους μικρούς γάδους και οι μικροί γάδοι που τους τρώει κάποιο άλλο ψάρι. Και οι πιγκουίνοι δεν τρώνε κάτι εκεί Τέλο πάντων, να αρχίσουμε τώρα και λέμε ποιο τρώει τι, ε, να, να μα πούνε και την άποψή του και οι επιστήμονε, αλλά τώρα δεν να πω. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή σταματήσουμε να λέμε όλα αυτά. Ε. είναι παράλογα. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Και ε, έναντι τη Επιτροπή και του Συμβουλίου να μην δεχθούμε τέτοιε μεθόδου. Ευχαριστούμε. Κύριε λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να παρακαλέσω ε, να παραμείνουμε επί της ουσίας σε αυτό το θέμα. Το να σχηριζόμαστε ότι εμείς ε, στην Ευρώπη ε, προσπαθούμε να λιεύσουμε με τρόπο που να μην καταστρέφει τα ψάρια, αυτό εντάξει το δέχομαι, αλλά από την άλλη βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε και απόλυτοι και τελείως θα χρειαζόμασταν μεταρρυθμίσεις. Πόρο απέχουμε από μια απόλυτα υγιή αλληλευτική πολιτική. Και θέλω να πω το στο σπίτι του πνιγμένου δεν δεν μιλάει κανείς για το σκηνή, του κρεμασμένου μάλλον. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι έχουμε μία συμφωνία ε, με την Ορβηγία και συμφωνήσαμε λοιπόν ότι το 85% της ε, του αποθέματο ε, που προτείνουν επιστήμονες μπορεί να είναι αντικείμενο αλίας. Το 15% ήταν ε, αυτό που απόμενε, το 10% ε, για την Ισλανδία και το 5% για τις νησφαιρόες. Αν λοιπόν τώρα προσθέσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε, βλέπουμε ότι οι δύο αυτές χώρες αλλιεύουν το 37%. Και αν προσθέσουμε το 85% και το 37% καταλαβαίνετε ότι έχουμε υπερβολική υπερ, υπεραλίευση. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Κατά την άποψή μου όμως ε, πρέπει να θεσπίσουμε και πράγματα που να είναι νομότυπα. Το να διαμαρτυρώμεθα. Ε, για το ότι η κυρία Δαμανάκη δεν διαμαρτύρεται, ε, αυτό το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω βεβαίως τους ε, αλληλείς που είναι αγανακτισμένοι, αλλά όχι και η Επίτροπος να επιβραβεύει τα παράνομα. Σας παρακαλώ να είμαστε περισσότερο επί της ουσίας. Γεγονός είναι λοιπόν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε και οι δικές μου πληροφορίες είναι οι εξή ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι διαπραγματεύσεις και υπάρχουν ελπίδες μέχρι τις 17 Οκτωβρίου περίπου, μέσα Οκτωβρίου, θα εξευρεθεί μια λύση. Εγώ προσβλέπω σε αυτό, προσβλέπω με την έννοια ότι περιμένω από την Ισλανδία ε, αν η Ισλανδία ενδιαφέρεται πράγματι να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να σέβεται τους δικούς μας τους κανόνες παιχνιδιού. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσαμε να οργανώσουμε κοινή ελληνική πολιτική και εδώ ανοίγω παρένθεση. Βεβαίως και υπολείπονται πάρα πολλά μέχρι του να μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά για την βιωσιμότητα και την αηφορία της Ισλανδίας. Και εδώ κλείνω την παρένθεση. Επανέρχομαι όμως στην Ισλανδία να μας πει αυτή πώς οργανώνει την πολιτική της τη ισχυρίζει ότι τα κάνει καλύτερα από εμάς. Προφανώς αυτό το λέω ε, χάρη ε, αστείου, αστείευόμενη. Πάντως, για μένα είναι παντελώς απαράδεκτο ένα κράτος μέλος να θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην τηρεί τους κανόνες αυτής. Τελειώνοντας, έχω και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δική της ε, την παρέμβαση άκουσα πάρα πολλά για αποθέματα ε, και θα ήθελα να ξέρω ε, σε άλλες διεθνείς διευθετήσεις τι ακριβώς συμβαίνει με τα ΤΑΚ. Η κατανομή των ποσοστώσεων πώς ακριβώς γίνεται. Νομίζω εδώ πρέπει να με βοηθήσει η Κομισιόν. Κατά τα άλλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε πιο επιστημονικοί, πιο αντικειμενικοί ε, στην ε, κουβέντα που κάνουμε και να στηρίξουμε την ε, Επίτροπο καλώντας την να λάβει μέτρα κατά της Ισλανδίας. Ευχαριστώ. Τα σχόλιά σας για τις Βρυξέλλες, τι να σας πω όσον αφορά ε, το 85% ε, του, ε, για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων ψαριών, όπως το προσφυγάκι, η υπεραλίευση γίνεται στα δικά μας τα νερά. Όμως υπενθυμίζω ότι όσον αφορά το σκουμπρί είναι πραγματικά τελεί, είναι, είναι πρωτοφανές κάτι τέτοιο. Φαίνεται λοιπόν φρικτό το γεγονός ότι εμείς υπονομεύουμε αυτή την, την ενιαία πιστοποίηση ε, επιτρέποντας τέτοιες συμπεριφορές από τις νήσους Φερόες και την Ισλανδία. Ίσως οι δύο ομιλητές θα ήθελαν να σχολιάσουν αυτά τα οποία άκουσαν. Και μετά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σπένσερ από την Επιτροπή. Ή θέλετε να ακούσετε πρώτα την Επιτροπή. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με όλα αυτά τα σχόλια των μελών της Επιτροπής Αλίας του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς πολύ συχνά ως κλάδος ε, μας, στη γωνία, μας στη γωνία και πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Και, και πολύ γενικά ε, η, ε, η κοινή γνώμη λέει «Μα κοιτάξτε τι έγινε και με τον τόνο The macro thing. Κοιτάξτε τι γίνεται και με τον ερυθρό τόνο. Ε, δεν μπορούμε, ε, είναι εύκολο να ε, στείλουμε τους ανθρώπους στη γωνία. Δεν λέω ότι ε, ε λιμένονται τους, τους πόρους μας έτσι μόνο, οι, μόνο Φερόες και η Ισλανδία. Απλά και μόνο λέω ότι εδώ μιλάμε για μια τακτική η οποία δεν βοηθά κανέναν. Κοιτάξτε, ε, ε, το ίδιο συμβαίνει και για με τη ρέγγα της ε, Βόρειας Θάλασσας. άρα λοιπόν όλα αυτά αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας μας. Αυτή η πολιτική είναι μέρος της φιλοσοφίας μας. Ε, μην παίρνετε τώρα ένα-ένα τα πράγματα ε, και μιλάτε για τα χέλια και για το προσφυγάκι. Ναι, το σκουμπρί είναι ξεχωριστό πρόβλημα και από μόνο το αποτελεί πρόβλημα. Όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Ρόντουστ, για την, ε, για την κλίδα κατανομής, πώς γίνεται η κατανομή των αποθεμάτων. Ε, δεν είναι ένα γραμμικό μέσο. Σας μίλησα ε, για την οτοκία, για την αναπαραγωγή, για την αύξηση των αποθεμάτων. Και σας είπα ότι θα γίνει αργότερα. Ε, γι' αυτό λέω να μην αφήσουμε την Ισλανδία να μπει στα δικά μας τα νερά. Εάν συμπεριλαμβάνουμε στην κατανομή προς την Ισλανδία και την πρόσβαση στα νερά μας, δηλαδή ανεξάρτητα με το μεριδιό του θα, θα, θα συνεχίσουν την αλία στα δικά μας τα νερά. Και αν ήμασταν πριν από λίγα χρόνια, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και να σας πω και το εξή. είναι ικανότατος ο στόλος τους. Αν υπήρχε σκουμπρί πριν το 2006, θα το είχαν βρει. Όπως και εμείς έτσι. Αλλά δεν υπήρχε τότε ε, στα νερά τους ε, σκουμπρί. Τώρα επεκτείνεται το είδος και έχουν σκουμπρί στα νερά τους. Γι' αυτό σας λέω μην τους αφήσουμε. Γιατί δεν γίνεται αναπαραγωγή εκεί. Τώρα, ε, τα πρόσφατα αλλιεύματα χρησιμοποιούνται για, την κατανομή των ποσοστώσεων. Και ακριβώς για αυτό το λόγο η Ισλανδία και οι νήσοι Φερόες προσπαθούν να αυξήσουν τα ολιευμά τους, γιατί ξέρουν ότι σε τελευταία ανάλυση, αν μιλήσουμε για κατανομή ποσοστώσεων, πολύ γρήγορα τα, θα μπουν και τα πρόσφατα επίπεδα λία στη συζήτηση. Αυτό δεν το θέλουμε εμείς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να αυξήσουμε ε, τα αλλιεύματά μας, γιατί έχουμε την πιστοποίηση, έχουμε τις άδειε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Και κάτι άλλο. Αν η Ισλανδία γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η ποσόστοσή τους ε, θα, ε, θα στηρίζεται ε, στα ιστορικά τους στοιχεία. Και αν μιλούν για 130.000 το χρόνο, καταλαβαίνετε πώς θα αυξηθούν αυτές οι επιδόσεις τους. Yes, thank you, Chairman. I Ο Ιαν Κάτ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολύ καλά τα συνόψω, ο συνάδελφος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις παρεμβάσεις τους. Και εγώ αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι δίνουμε, ε, δίνετε εσεί μάλλον στην Επιτροπή Ελληνία ε, ένα ισχυρό μήνυμα. Ότι θα έχουμε μια αποσασιστική στάση απέναντι στα νησιά Φερόε και την Ισλανδία και δεν θα επιβραβεύσουμε την ανεύθυνη στάση του. Για το απόθεμα, μια ερώτηση. Γιατί είναι τόσο, ήταν κατά το παρελθόν τόσο επιτυχημένο το απόθεμα. Η συνταγή είναι απλούστατη. Χρειάζονται καλές επιστημονικές συμβουλές, ένα σχέδιο διαχείρισης που θα τηρείται και αυτό το οποίο όλα αυτά τα βελτιώνει είναι να τηρούνται και οι όροι των ε, λευτικών συμφωνιών. Αν δεν υπήρχαν αυτά, αυτοί οι παράγοντες, ε, θα υπήρχαν προβλήματα και θα υπάρξουν προβλήματα. Θέλω λοιπόν για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας και να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι οι λευτικές μας κοινότητες δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρί αλληλευτικά δικαιώματα. Έχουμε την καλύτερη, τον καλύτερο στόλο και τι καλύτερε υποδομέ. Αν δεν έχουμε δικαιώματα, τι να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να βγούμε στη θάλασσα να ψαρέψουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στον άνθρωπο ο οποίο ε, έχει την πολύ δύσκολη δουλειά όλε αυτέ τι φιλοδοξίε να τι κάνει πραγματικότητα στι διαπραγματεύσει με τα παρακτέα κράτη, με την Ισλανδία, με τα νησιά Φερό. Από την Επιτροπή λοιπόν τον λόγο έχει ο κύριος Σπένσερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Προσεκτικά άκουσα τις πολύ καλές παρουσιάσεις ε, των κύριων Μπάλσφορτ και Γκάτ. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την απογοήτευσή τους για τις, απο... εξελίξεις που είχαμε κατά το έτος 2010. Και εμείς ξέρετε ε, πώς, έχουμε αξιολογήσει την μονομερή ποσόστοση των Φερόε και, το, και της Ισλανδίας, που είναι απαράδεκτη τα επίπεδα, δεν βασίζονται ούτε σε κάποιο αρχείο, σε κάποιο ιστορικό, ούτε και στις επιστημονικές συμβουλές. Και όπως υπόθηκε νωρίτερα στην παρουσίαση, οι δράσεις των δύο αυτών κρατών είναι πραγματικά καιροσκοπικές, που την έννοια ότι εκμεταλλεύονται την αύξηση, την αυθονία του αποθέματος, που βέβαια κατέστη δυνατή και φυσικά χάρη στις προσπάθειες τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία με την κοινή διαχείριση των αποθεμάτων που ακολουθούν τα τελευταία δέκα χρόνια. Τώρα, το είδο των δράσεων που ε, στις οποίες προβαίνουν η Ισλανδία και τα Φερόε ε, ε, σίγουρα υπονομεύει την βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Και αυτή είναι η πρώτη στη ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βιωσιμότητα των αποθεμάτων μας ενδιαφέρει, διότι με τέτοια υψηλά επίπεδα ακούσαμε να γίνεται αναφορά σε 930.000 τόνους αλλιεύματα για φέτος που υπερβαίνει κατά πολύ το ΤΑΚ των 570.000. Θα δούμε τι θα γίνει το 11, αλλά είναι, ε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μειωθούν τα αποθέματα. Και είχαμε πολύ κακές ε, εμπειρίες που θα επαναληφθούν με το προσφυγάκι και το απόθεμα που χωρίς καμία συμφωνία ανταλλαγής ε, τα πήγαινε καλά ως απόθεμα και όταν υπήρξε συμφωνία τα πράγματα πλέον είχαν φτάσει στο ως εδώ και μη παρέκει και τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου η σύσταση ΤΑΚ για το προσφυγάκι θεωρείται ως πάρα πολύ χαμηλή για του χρόνου. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε την ίδια ιστορία λοιπόν, ούτε θέλουμε να απειληθεί η βιωσιμότητα, άρα μείωση των αλληλευτικών δυνατοτήτων. Και αυτό δεν το θέλουμε γιατί θα έχει άμεση επίπτωση ε, στον βασικό εμπλεκόμενο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ισπανία, στο Βισκαϊκό και στη Βορεια Θάλασσα ε, γεννούν τα αυγά τους αυτά τα ψάρια και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι μόνο ε, εκεί, είναι κοινοτικό αν θέλετε ψάρι αυτό. και λίγη οτοκία βλέπουμε και στην Ισλανδία και στα Φερόε αυτόν τον καιρό. Τώρα, πρέπει να λάβουμε βέβαια υπόψη και τι κινήσει, τη μετακίνηση των αποθεμάτων. Να δεχθούμε ότι υπήρξε μετακίνηση, γι' αυτό και τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 100.000 τόνους μπόρεσαν να ληφθούν ε, στην Ισλανδία. Το 23% του ΤΑΚ που συνιστάται. θα έχουμε κάποιες ιδέες ε, για την αλία του 2011 πώς θα πρέπει να διεξάγεται για την Ισλανδία. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τα στοιχεία. Αλλά ο στόχος μας βέβαια είναι να έχουμε συμφωνία και με τα τέσσερα παράκτια κράτη. Όλοι μαζί να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι ο στόχο τη Κομισιόν και τη Ένωση. Και θέλουμε μια μακροπρόθεσμα ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείριση ε, και ανταλλαγή ώστε να έχει ο κλάδος την απαιτούμενη σταθερότητα. Αναζητούμε λοιπόν την επίτευξη συμφωνία. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω όμω και ήταν σαφέ το μήνυμα και του Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα. Δεν θέλουμε μια συμφωνία με κάθε τίμημα, με οποιοδήποτε τίμημα, για του για τους λόγου που αναφέρατε κι εσεί. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλουμε να επιβραβεύσουμε αυτό το οποίο εμεί θεωρούμε ανεύθυνη αλληλεία. Ε, εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί οι συμβαλόμενοι και να είναι και υπεύθυνοι στις ενεργειές τους. Ούτε υπεύθυνο είναι ούτε ρεαλιστικό. Συμβαλόμενα μέρη όπως η Ισλανδία και τα Φερόε να βγάζουν ε, από το κεφάλι τους ε, αριθμητικά στοιχεία όπως το 23%. που πού προήλθε αυτό το 23%? Παίρνει το ποσοστό και το συγκρίνει ε, με το ποσοστό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται έτσι η κατανομή. Το ίδιο με τα Φερόε είπαν πέρυσι ότι θέλαν αύξηση. Τι θέλετε, τους είπαμε εμείς. 15% μας είπαν. Μα δεν μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί με αυτή τη βάση. Πρέπει να είναι σωστή η βάση διαπραγμάτευση. Να υπάρχει και κάποια στήριξη, επιστημονικά στοιχεία στα οποία να βασιστεί κανείς. Αυτό που είπε η κυρία Ροντάστ τι στοιχεία ε, χρησιμοποιούνται για την πολισμό της κατανομής, για την κλίδα κατανομής. Είναι τα επίπεδα αλλιευμάτων, ε, η συμβολή στο απόθεμα λόγω παραδοσχάρη εκτροφής και τα κτλ. Ε, περιβαλλοντικός έλεγχος. Τι ακριβώς λένε τα ΦΕΡΟΕ, πώς θα αποδείξουμε θα μπορούσαμε να είχαμε αλλιεύσει περισσότερα ψάρια τα τελευταία δέκα χρόνια. Είμαστε μέσα στη συμφωνία ε, παράκτιων κρατών που περιορίζεται τις αλληλευτικέ μας δυνατότητε θα πούν. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όταν βγάζει έτσι, όπως ε, στα κουτουρού, όπως της έρχεται η Ισλανδία ένα νούμερο στον αέρα, μας δημιουργεί προβλήματα. Και όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία, όχι όμως όποια να είναι συμφωνία. Και πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του ελευτικού κλάδου προς την κατεύθυνση αυτή, προς μια υπεύθυνη δηλαδή προσέγγιση στη διαχείριση. Η διαβούλευση στο Συμβούλιο ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου. Ο στόχος μας ήταν να τους δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την δραστηριότητά τους και θέλουμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Ε, δεν ήταν διαπραγματεύσεις, ήταν συζητήσεις, αλλά ήταν ένα προήμιο των διαπραγματεύσεων για να καταλάβουν τη θέση μας και να καταλάβουμε εμεί και από πού έρχονται. Όσο επίσης σημαντικός εμπλεκόμενος και η Νορβηγία θα έχει συζητήσει και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθυντών από αυτήν την εβδομάδα και θα υπάρχουν τεχνικέ συζητήσει με την Νορβηγία πριν από τι διαπραγματεύσει του Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί έχουμε τη συμφωνία με την Νορβηγία πρώτα απ' όλα. Να μοιραστούμε τι θυσίε που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτή τη συμφωνία των κρατών. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι συμφέρει πάρα πολύ και τι δύο πλευρέ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νορβηγία. να τακτοποιήσουμε τα πράγματα με την αλήθεια αυτή. Τέλος, αυτό το οποίο θα μπορούσα να σας προτείνω είναι το εξής. Όπως έχει κατάσταση, είναι πολύπλοκες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αν θέλουμε να καταλήξουμε σε εξισορρόπηση των διαφόρων συμφερόντων και θα χρειαστεί κατά την άποψή μου να γίνουν πολλές συναντήσεις. Μία από αυτές τις συναντήσεις διερευνητικά την ε, έχουμε προγραμματίσει στα τέλη Οκτωβρίου που λέτε εσείς να κάνετε τη δική σας ακρόαση, κύριε Πρόεδρε. Εδώ δεν ξέρω αν λοιπόν θα είναι εφικτό. Θα είναι μάλλον δύσκολε οι διαπραγματεύσει. Θα σα κρατούμε ενήμερου ε, για τι εξέλιξει όλη τη διάρκεια αυτού του εγχειρήματο. Και τώρα, αν με επιτρέπετε συντομία, θα ήθελα να σχολιάσω τι παρεμβάσει των βουλευτών τη Επιτροπή σα. μπορώ να σας καθησυχάσω ότι το θέμα του σκουμπρίου είναι προτεραιότητα στις παρεμβάσεις μας για την Ισλανδία. Και μιλώ για το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Και επίσης ε, η σας ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αυτό που υποσιαστικά ήταν, ε, δεν θεωρούμε το χρονοδιάγραμμα το ενταξιακό να είναι το ίδιο με την μακροδιαχείριση του σκουμπριού οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει μπορούν να συνεχίζονται. Εμεί θέλουμε τώρα για το σκουμπρί, όχι μετά από <laughs> χρόνια να καταλήξουμε κάπου. Φυσικά, σαν υποψήφια χώρα ε, για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισλανδία θα πρέπει, είναι σαφέ αυτό, να έχει μια συμπεριφορά που θα σέβεται το κεκτημένο τη Ένωση. Και αυτή η ελεύθερη αλή από το 2007 που είχε η Ισλανδία δεν θα επιτραπεί στο πλαίσιο της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, είτε ως έχει τώρα, είτε όπως θα προκύψει μετά από το 2012. Δεν θέλω τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες για τις ποσοστώσεις ε, των ε, νησιών Φερό όπως έχουν αυτή τη στιγμή. η κακήρωση της ποσόστασης αυτής όπως ακυρώνει και τις ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη για το 2010 σε διμερές επίπεδο με τα αφαιρό. Και αυτό αφορά αρκετά διαφορετικά ε, αποθέματα που ενδιαφέρουν αρκετά κράτη-μέλη. Στο Συμβούλιο ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε ομοφωνία. Αν και δεν συζητήθηκε βέβαια με λεπτομέρεια. Όπως είπα λοιπόν, εστιάζουμε στο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία Σαφώς όμως έχουμε πει, το έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκάθαρα, ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, εάν οι προσδοκίες της Ισλανδίας και των Φερόε για τις ποσοστό, εξακολουθήσουν να είναι ανεδαφικές σε ό,τι αφορά το επίπεδο, ε, θα λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν το τέλος ε, του έτους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντως ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Uh, Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, πολύ περιεκτική, ουσιαστική η παρέμβασή σας. Να διαβάσετε τις ευχαριστήσεις μας και στην Επίτροπο, στην κυρία Δαμανάκη. Γιατί και αυτή έδειξε έτσι σθένος στην αντιμετώπιση όλων αυτών των εξελίξεων. Και κάτι άλλο που ο κ. Βαν Μπέλσεν σχολίασε ότι οι Φερόες ε, μέσα αυτή τη νέα συμφωνία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας ε, και αναφέρεται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εισακούεται και ελπίζω στο μέλλον αν υπάρξουν νέες συμφωνίες που θα τεθούν στη σκή, θα ενημερωθούμε και εμείς πλήρως. Με το βάση το άρθρο 218, παράγραφος 6, η Κομισιόν πρέπει να μας ενημερώσει και να ακούσει την άποψή μας. Αυτό είναι το παιχνίδι, με αυτούς τους κανόνες παίζεται πλέον. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ε, καταλήξουμε με έναν ικανοποιητικό συμβασμό που θα ωφελήσει όλους. Και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι τα διάφορα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος που θέλει να θίξει κάτι στα διάφορα. Αν όχι, 16 ανακοινώσει του Πρόεδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Νομίζω η Γραμματεία έχει ε, μοιράσει το έγγραφο με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Η ημερομηνία διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 26 Οκτωβρίου Θα συναντηθούμε και θα είναι και η κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε και θα τα πούμε στο Στρασβούργο.